Καλημέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ. Πάρτε θέσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ανακοινώσω ότι πρέπει να έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Ετοιμάστε τις παρακαλώ. Βάλτε τις στο μηχάνημα. Όσοι το έχουν ξεχάσει, πείτε να σας τις φέρουν, διότι έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα το πρωί, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ανακοινώσω τι θα, τίνος πράγματος θα ψηφίσουμε, αλλά να σας θυμίσω ότι στη συνέχεια, όπως και χθες, ε, έχουμε πολύ φορτωμένη σε διάταξη μια σειρά από εκθέσεις υπηρεσιών ε, για ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα έρθει και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς εδώ στην Επιτροπή μας. Οπότε πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, διότι η παρουσίαση του κυρίου Τίμερμαντς είναι να ξεκινήσει 9.45. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Ξεκινούμε λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία για δύο φακέλους που έχουν να κάνουν ε, με τη χρηματοδότηση για το έτος 2020, τον προπολογισμό, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω ο κύριος ε, Ραρό έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα απλώς να κάνω μια, ένα σχόλιο, λέει ο Γκαρό. Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξεπλάγην που δεν είναι μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες ε, δεν είναι μεταφρασμένα όλα τα κείμενα από τα οποία ε, θα ψηφίσουμε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες που προφανώς λόγω κατεπήγοντος τα λαμβάνουμε μόνο στα αγγλικά, αλλά το κείμενο, το αρχικό κείμενο με το οποίο ψηφίζουμε θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο. Το λέει ο κανονισμός, το άρθρο 169 που λέει ότι οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μόνο έχουν, ε, αφόσον έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Το αρχικό κείμενο τουλάχιστον ε, των τροπολογιών θα έπρεπε να ε, έχει μεταφραστεί. Δεν είμαι λοιπόν σε θέση ούτε εγώ ούτε και άλλοι να πάρουμε θέση για ένα σημαντικό κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία. Δεν, είμαι, δεν μπορώ στην πραγματικότητα να ψηφίσω το οτιδήποτε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας κύριε Γκαρό, τα σημειώσαμε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση αυτή είναι πραγματικά εξαιρετική. Είμαστε στην αρχή της περίοδου των εργασιών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, μια μεταβατική φάση λοιπόν, και είπαμε ότι υπάρχει πίεση χρόνου. Πήραμε την απόφαση στην ομάδα του συντονισμού λόγω της πίεσης χρόνου ε, να προχωρήσουμε έτσι να γίνει δηλαδή αυτή η ψηφοφορία τώρα επειδή υπάρχει πίεση χρόνου και γι' αυτό δεν υπάρχει μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό. Πρόκειται για μια εξαίρεση. Ε, σας ζητώ συγγνώμη συνήθως ε, υπάρχει η, διαδικασία γίνεται σεβαστή μάλλον και τα κείμενα υπάρχουν σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Και εσείς επί της διαδικασίας δεν μπορούν να αλλάζουν ε, τον κανονισμό οι συντονιστέ. Αν λέει ο κανονισμό ότι πρέπει να είναι διαθέσιμε οι μεταφράσει σε όλε τι γλώσσε, δεν μπορούν ε, να είναι υπεράνω του κανονισμού οι συντονιστές. Ναι, εντάξει, ακούστε. Η απόφαση πάρθη από την Επιτροπή των Συντονιστών. Οπότε τώρα οφείλουμε να προχωρήσουμε. Σε παραλαμβάνω, 9 από τα θα έρθει ο κύριο Τίμερμαν, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία λοιπόν. Σημείο 12 τη ημερήσια διάταξη. Γενικό Προπολογισμό ε, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Έχουμε δύο ψηφοφορίε και οι δύο αποτελούν εκθέσει τη ε, συναδέλφου Γκουέντολιν Ντέλμπο Κόρφιλντ. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του σχεδίου ε, γνωμοδότησης και στη συνέχεια ε, ψηφίζουμε και επί των τροπολογιών. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σχέδιο γνωμοδότησης, έτσι. Συμβασμός 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός, ε, ε, μάλλον τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ε, 13, συγγνώμη. Τροπολογία 13, διορθώνει ο πρόεδρο. Ναι, λίγο πιο αργά παρακαλώ. Είμαι νέο μέλος, ε, προσπαθώ να παρακολουθώ και τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Τροπολογία 13, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Βλέπετε ότι είναι 29-29, αλλά όταν υπάρχει ισοψηφία απορρίπτεται. Χρειάζονται περισσότερο θετική από αρνητική ψήφους. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία 34 αν δεν κάνω λάθος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. 48, έτσι. 48. Είναι η σελίδα 5 του καταλόγου. Τροπολογία 48. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έγινε ένα τεχνικό λάθος, θα πρέπει να επαναληφθεί αυτή η ψηφοφορία, συγγνώμη. 53 λοιπόν εκ νέου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ιντεβέλτ. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβασμός 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβι... Ε, συγγνώμη, τροπολογία 60. Υπε... Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Απορρίπτεται. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 64. Στην τελευταία σελίδα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Από ό,τι μου λένε υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ που περισσεύει εδώ. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 66 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίσουμε το συνόλου του κειμένου όπως τραγωποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται να συγχαρούμε την κυρία Ντελμπό Κολφίλτ για το έργο της. Και τώρα περνάμε στις τροπολογίες Εδώ έχουμε πιο μακρύ κατάλογο ψηφοφορίας, γι' αυτό πρέπει να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή. Ξεκινούμε λοιπόν με την έκθεση της ίδιας συναδέλφου Κουέντολιν Τελμπο Κόρφιλτ, δημοσιονομικές ε, τροπολογίες για τον προϋπολογισμό 2020. Ξεκινούμε λοιπόν. Τροπολογία 5809 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-45. Άρχεται ψηφοφορία. 58.45. έτσι. Πέρασε ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τώρα 58-46. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-47. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-36. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58-17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 58-34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58-35. Άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβιβαστική 3 όχι τι πρέπει να την ψηφίσουμε α συγγνώμη ξέχασα την 58-19. άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε και τώρα συμβιβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση. εγκρίνεται. Τροπολογία Τροπολογία 58-20. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5833. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 58-48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 58-81. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 58-39 άρχεται η ψηφοφορια περασε Πέρας. Εγκρίνεται. 58-52 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-03. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε. Α, είναι κάποιες ταυτόσιμες τροπολογίες προς αυτή που μόλις εγκρίναμε. Άρα πηγαίνουμε στην 5805, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 58-57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 58-58. Άρχεται. Πέρας. 58-59. 58-59, 58-59, αρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 58-25, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58-60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 58-42 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 5843, 58-43 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58, 28, 58, 63 Άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρας. Εγκρίνονται 58-00. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 58-11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-29 και 58-64 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Προφορική τροπολογία 58-83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-10. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 58-80. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-04. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-12 και 58-65 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνονται. 58-13 και 58-66 ταυτόσημες άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 58-14, 58-67 ταυτόσημες άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται 58, 15 και 58, 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται και 58, 16, 58, 69 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. Προχωρούμε. Προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία. Ελέγχουμε ονομαστικά το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Τη συνάδελφο. Κοιτάξτε που μας μείνανε και λίγα λεπτά διάλειμμα. Σε ένα τέταρτο θα έρθει ο κύριος Τίμερμανς. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας λοιπόν και θα είμαστε έτοιμοι εδώ στις 9.45 για να ακούσουμε τον κύριο Τίμερμανς.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 Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε ήσυχω. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας και μάλιστα στην ώρα μας. Ας καλωσορίσουμε θερμό τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν. Είναι τιμή μας να τον ακούμε Πάντοτε εκτιμούσαμε τον πρόσφατο διάλογο που είχαμε σε όλη την προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και συνολικώς του Ευρωκοινοβουλίου. με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα που άπτονται τα νομοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Υπήρξαν και άλλοι επίτροποι, αλλά εσεί είστε το καθήλυνα αρμόδιο, κύριε Τίμερμαν. Σα έχουμε συνηθίσει εδώ. Θέλουμε λοιπόν να ενημερωθούμε για θέματα κράτους δικαίου. Ένα από τα βασικά ζητήματα που είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες ένα θέμα προς συζήτηση ιδιαίτερα επικαιρό και σημαντικό. Είδαμε το συνταγματικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κανόνων και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Μα ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των κοινοβουλίων και του κοινοβουλίου, μα ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των πολιτών, το κράτο δικαίου, η δημοκρατία. Μα ενδιαφέρουν οι αρχέ και οι αξίε που καταγράφονται στι συνθήκε και στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 εγγράφεται το δικαίωμα, ε, μάλλον το, το τι είναι το κράτος δικαίου ορισμός. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αντιπρόεδρο Τίμερμανς, ο οποίος μόλις πρόσφατα πέτυχε να υπάρξουν αποτελέσματα σε δύο περιπτώσεις, δύο επεισόδια του Απριλίου και του Ιουλίου 2019, με δύο έγγραφα. Έγγραφα για την ενίσχυση του πλαισίου κράτους δικαίου βάσει τη σύσταση και αυτή τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό πρόληψη σε αυτόν τον τομέα. Δημοκρατία, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Σκοπός είναι να καλυφθούν κάποια κενά και να διορθωθούν κάποιες διαδικασίες βάσει της διατύπωσης του άρθρου 7 ως τώρα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε όλοι τα τελευταία συμβάντα των τελευταίων ετών τα οποία χρειάστηκε να βιώσουμε. Έχουμε λοιπόν ένα αποτύπωμα για τη δράση μας στο μέλλον, ε, Ιούλιος 2019, 17 Ιουλίου, με τίτλο Ενίσχυση του πλαισίου κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντιπρόεδρο Τίμπρεμαν θα μα το αναλύσει και θα συζητήσουμε. Σίγουρα υπάρχουν πολλέ προσδοκίε. Οπότε να ε, παρακολουθήσουμε και το πόσο χρόνο έχουμε. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων με τους συντονιστές. Μετά θα δώσουμε το λόγο στα μέλη που τον επιθυμούν. Αλλά σας προσκαλώ γιατί έχουμε μια μισή μόλι ώρα, 90 λεπτά στη διάθεσή μα και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολλοί άριθμοι συνάδελφοι που θα σηκώσουν τα χέρια τη κάρτες του, παρακαλώ περιορίστε τη διάρκεια τη παρέμβασή σα σε ένα λεπτό ακριβώ. ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε, Φράν. Πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για, την για το ευγενικό καλωσόρισμα. Πολλά τα οικεία πρόσωπα, αλλά και πολλά τα νέα που ελπίζω ότι θα γίνουν οικεία σύντομα και ότι θα γνωριστούμε καλύτερα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Η Ευρώπη χρειάζεται το Ευρωκοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και όλοι μαζί πρέπει να βρούμε απαντήσεις στις απορίες και τις ανάγκες των πολιτών. Σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσω για την ανακοίνωση που έχει να κάνει με την ενίσχυση του πλαισίου κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανακοίνωση που εγκρίναμε τον Ιούλιο. Το ευρωπαϊκό μα εγχείρημα βασίζεται στον διαρκή σεβασμό του κράτου δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι προπόθεση για να λειτουργεί η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και για την ε, πραγματική εφαρμογή του κράτου δικαίου, την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά και για το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον οι απειλέ κατά του κράτου δικαίου ε, αγγίζουν την καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια και απειλούν τι ε, αξίε και την ταυτότητά μα, ε, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι 89% όσων ερωτήθησαν απαντούν ότι το κράτο δικαίου και ο σεβασμό του κράτου δικαίου είναι ουσιαστική σημασία όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλα εκτός Ένωσης, στην Ευρώπη γενικώ. Είναι κοινή ευθύνη λοιπόν των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και όλων των πολιτών. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και αυτήν την Επιτροπή για τη δέσμευσή της σε αυτόν τον ε, χώρο. Ένας από τους σκοπούς της ανακοίνωσης που εγκρίναμε τον Ιούλιο είναι να ξεκινήσουμε από το τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να υπάρχει μια καλύτερα συντονισμένη διαθεσμική προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί το κράτο δικαίου στην Ένωση. Η ανακοίνωση βασίζεται στη διαδικασία ε, μελέτη που ξεκίνησε τον Απρίλιο και λαμβάνει υπόψη τι προτάσει σα για τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις αξίες και το κατός δικαίου ε, με τις συστάσεις που συνέταξε η Επιτροπή σας, καθώς και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την εμπειρία της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια σειρά από συγκεκριμένε δράσεις ε, σε τρεις βασικούς τομείς. Πρόθεση, πρόληψη και ε, απάντηση. Η πρόθεση έχει να κάνει με την δημιουργία προτύπων βάσει της νομολογίας και μια κοινή κουλτούρα κράτους δικαίου. Η πρόληψη έχει να κάνει με την έγκαιρη ανείχνευση των προβλημάτων κράτους δικαίου, ώστε να μην διωγωθούν περαιτέρω και να υπάρξει υποστήριξη για την ανίσχυση του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίω. Προτιμούμε την πρόληψη από την ανάγκη αντίδρασης. Όμως και η αντίδραση απαιτείται. Πρέπει να ενισχύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους εθνικούς μηχανισμούς που δεν είναι εύρωστοι. Εδώ και στου τρει πυλώνε, το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο. Ξεκινώντα από την πρόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχύσουμε το κάτω δικαίου και τη σχετική κουλτούρα σε όλο το γενικό κοινό. Πρέπει να υπάρχουν καλύτερε ε, γνώσει για τι ε, απαιτήσει του κράτου δικαίου και τα πρότυπα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιοποιήσει όλε τι δυνατότητε χρηματοδότηση για να επιτρέψει στου ενδιαφερομένου, ε, ιδίω τη κοινωνία των πολιτών, να μάθουν περισσότερα. Με ετήσια εκδήλωση για το κράτο δικαίου που θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι από την κοινωνία των πολιτών και τι οργανώσει των πολιτών. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την κοινή μα κληρονομιά, τι κοινέ μα αξίε. Ε, όταν υπάρχουν απειλέ ή επιθέσεις ή ε, αναταραχέ που έχουν να κάνουν με το κάτω δικαίου στην κοινωνία των πολιτών, πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση. Και τα εθνικά κοινοβούλια, οι βουλέ έχουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Γι' αυτό, βάσει των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να καταρτήσουν ε, μορφέ συνεργασία και κοινοβουλευτικέ για το κράτο δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεισφέρει και να υποστηρίξει. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει το πλέον καινοτόμο στοιχείο τη ανακοίνωση, δηλαδή τη δημιουργία μια ετήσιας, ενός ετήσιου κύκλου αναθεώρησης για τα θέματα κατ' δικαίου. Αυτό βασίζεται στην αναγνώριση ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα εντοπισμού προβλημάτων στα κράτη-μέλη τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες με το κάτω δικαίου και να προτείνουμε πιθανές λύσεις. Πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την έννοια και γι' αυτό θα παρακολουθούμε στενότερα το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Προτείνουμε να οδηγηθούμε στην ενίσχυση τη διαθεσμική συνεργασία για το θέμα αυτό. Γνωρίζω ότι είναι κάτι που ζητά το Ευρωκοινοβούλιο ε, χειρά και ε, με επιμονή εδώ και καιρό. Θα πρέπει λοιπόν στα κάτι που υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ε, ιδίω προβλήματα δρόμηση, να, ληφθεί, ε, να αναλυθεί δράση. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε μάλιστα ε, με τον κύκλο αυτό το τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία θα ετοιμάζουμε και μια ετήσια έκθεση για το κράτο δικαίου, για τι περαιτέρω εξελίξει και ίσω και ένα βαθμολόγιο. Η ετήσια έκθεση θα παρουσιάζει μια συνοπτική επισκόπηση για τι εξελίξει, αρνητικέ ή όχι, στα διάφορα μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό, και για το κράτο δικαίου, το τι συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και άλλε πληροφορίε. Η έκθεση θα χρησιμοποιείται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ω βάση για τι συζητήσει του. Και λίγα λόγια για δύο σημεία που γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντο για την Επιτροπή σα. Πρώτα απ' όλα το πεδίο τη παρακολούθηση και η ανεξάρτητοι πυρογνώμονε. Για το πεδίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του κράτου δικαίου. Αυτό όμω έχει και επιπτώσει στην δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι προπόθεση το κράτο δικαίου για την προστασία τη δημοκρατία και των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμω πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η δικαστική προστασία, καθώ και αυτή και ο σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι από τι βασικέ συνιστώσει του κράτου δικαίου. Γι' αυτό οι αξίε αυτέ είναι αλληλένδετε, στενά συνδεδεμένε με το κράτο δικαίου. Πρέπει λοιπόν, εφόσον προστατεύουμε το κράτο δικαίου, να αποδεχτούμε ότι προστατεύεται και η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίση, η ανακοίνωση εξηγεί ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν στην καταπολέμηση τη διαφθορά και αυτή καλύπτεται. Σχετίζεται με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όλο αυτό. Ε, η πολυφωνία στα μέσα μαζική ενημέρωση και ελεύθερε εκλογέ είναι κομμάτι τη ίδια προσπάθεια. Θα πρέπει βεβαίω τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία ε, να μην τα εγκαταλείψουμε στην τύχη του. Οι θεμελιώδει αξίε μα απασχολούν εξίσου και γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε το σεβασμό του και την τήρησή του. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, καταγράφουμε τον σεβασμό του από τι χάρτε και τι εκθέσει των κρατών μελών και σκοπεύουμε να καταρτήσουμε μια συνοπτική ε, χάρτα. Θέλουμε να δούμε το επίπεδο της επιβολής ε, λόγω χάρη παρακολουθούντα στενότερα την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, το Σεπτέμβριο του 2018 ε, εγκρίναμε ένα συνολικό πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την προστασία τη δημοκρατία και τη διοργάνωση ανεξάρτητων και ελεύθερων εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ξέρετε ότι η πρόεδρο Φοντερ Λάιεν έχει αναλάβει τη δέσμευση να εγκρίνει κατευθυντήριε γραμμέ και μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση τη δημοκρατία. Για τι ανεξάρτητε εκλογέ. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο πρότεινε τη δημιουργία πάνελ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που να αξιολογούν την κατάσταση και να σφιγμομετρούν το τι συμβαίνει στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη. Παρά την ένδειξη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ίσω δημιουργεί το, μια σειρά από προβλήματα ω προ την νομιμοποίηση, της, ε, την εξισορρόπηση των συνεισφορών των ΜΕΝ και των ΔΕ και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Πάντω, αξιοποιούμε όλε τι πηγέ εμπειρογνωμοσύνη και ε, κοιτάζουμε να τι τι πληροφορίε μα, γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε προγνωμοσύνη τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να εκπορεύεται από εμά αυτή η αξιολόγηση. Ιδίω όταν η δράση που προτείνουμε έχει νομικέ και οικονομικέ συνέπειε. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία ε, τη πηγή ε, τη προγνωμοσύνη μα, όπω τη Επιτροπή τη Βενετία, των δικτύων ε, νομικών εμπειρογνωμόνων, τη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά. Για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Η Επιτροπή τη Βενετία, λόγω χάρη, είναι αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο τη προσοχή μα και επηρεάζει όσα κάνουμε. Στον τρίτο πυλώνα, την αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την ε, δεσμευσή τη να παραμένει θεματοφύλακα των συνθήκων. Ε, υπ' αυτήν την έννοια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογράμμισε του τελευταίου μήνε με ε, μοναδικέ αποφάσει του τη σημασία του δικαστικού τομέα στην εύρωστη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιζόμενοι σε αυτή την ομολογία, θα αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για τι διάφορε δικαστικέ διαδικασίε. Η ε, αποτελεσματικότητα των ε, διαδικασιών φάνηκαν και στην περίπτωση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας με μια απόφαση που το αφορά και ήταν ιστορική. Εκεί το δικαστήριο αποφάσισε ότι η πολωνική νομοθεσία που αφορά τη μείωση της ηλικίας συνταξιδότησης όπως εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολωνίας αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και παραβιάζει την αρχή της ε, μη δυνατότητας, μάλλον της, της απαγόρευσης μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών. Ε, και της λήψης απόφασης από αυτούς. Ε, άλλες διαδικασίες επί παραβάση ε, εκκρεμούν και στις 17 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει απάντηση από τις πολωνικές αρχές για την πρόσφατη γνωμοδότηση που έχει να κάνει με το πειθαρχικό καταστατικό των Πολωνών Δικαστικών Υπουργών καθώς και της ηλικία συνταξιοδότηση, του ορίου συνταξιοδότησης των τακτικών δικαστικών λειτουργών στα πολωνικά δικαστήρια. Υπάρχει επίσης διαδικασία επιπαραβάσης κατά της Ουγγαρίας, που έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης της, κοινων... διοργάνωσης των οργανώσεων τη κοινωνίας των πολιτών και της μεταχείρισης των ετούντων ασύλου. Εδώ ε, ε, οι υποθέσει αυτέ εκκρεμούν ακόμα ενώπιον του δικαστηρίου όσο προ την διαδικασία του άρθρου 7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στην ε, ανακοίνωσή του να εντείνουν τη συλλογική του προσέγγιση. Η ανακοίνωση το τονίζει, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει απαραίτητη θεσμική ισορροπία στο Κοινοβούλιο και ότι μπορεί με τη διαδικασία του άρθρου 7 το Κοινοβούλιο να προβάλλει τα επιχειρήματά του. Αυτό ξεκίνησε σε επίπεδο Συμβουλίου και ενθαρρύνουμε το, τα δύο θεσμικά όργανα να εγκρίνουν σύντομα ε, την, τον κανονισμό για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε τι διαρκεί ελλείψεις ό,τι αφορά το συμβασμό κατ' δικαίου από τα κάτι μέλη. Πιστεύω ότι είναι ένα ε, απαραίτητο εργαλείο για να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εν είδη συμπεράσματο, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανυπομονεί τους ερχόμενους μήνες να έχουμε έναν καρποφόρο και πλούσιο διάλογο με όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κάτι μέλη για ένα ισχυρότερο, καλύτερο πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σα έχει διδαματίσει σοβαρό ρόλο τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι αυτό τον κέριο ρόλο θα συνεχίζετε να τον φέρετε ει πέρα σε πάξη έω ε, το τέλο τη θητεία. Έχουμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε μπροστά μα και πιστεύω ότι μαζί, χέρι-χέρι, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε την Ευρώπη πιο ελεύθερη, πιο δυνατή. Οι πολίτες μας να αισθάνονται ότι το κάτω δικαίωμα τους προστατεύει ό,τι και αν συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε, για τη σύντομη αυτή παρουσίαση του τελευταίου έγγραφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό. Πολύ σωστά είπατε εδώ και καιρό το ζητάει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Από το 2016 τουλάχιστον, ε, στα ψηφίσματά μας ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει αυτό τον μηχανισμό, τον προληπτικό για το κράτος δικαίου που θα περιλαμβάνει όλα τα συστατικά ε, ε του τι είναι κράτος δικαίου για μας ε, τους Ευρωπαίους σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα πεδίο συζήτησης. Ε, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μιλητών. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστέ. όμως σα παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Δύο λεπτά και μετά ένα λεπτό. Όσοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα, να τα γράψετε ενδεχομένως. Για να μπορείτε όντω να τα πείτε σε ένα λεπτό. Ξεκινούμε με τους συντονιστές από το ΕΛΚ Πρώτα, η κυρία Ματσόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Αντιπρόεδρε, που μας παρουσιάσατε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μία ένωση κοινών αξιών και γι' αυτό καλωσορίζουμε αυτήν την ανακοίνωση της Κομισιόν του Ιουλίου. Είναι ένα βήμα για να εξασφαλίσουμε ότι το κράτος δικαίου θα γίνει σεβαστό σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Όπως μόλις είπατε, θα πρέπει αυτή η ανακοίνωση από εκεί πέρα να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε δράσει και μέτρα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ελευθερία τύπου, ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Creative Europe, ε, στα πλαίσια του προγράμματο αξιών, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα τα ανεξάρτητο τύπο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Όμω πρέπει να πάμε πέρα από τη χρηματοδότηση και να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε την πίεση που δυστυχώ αυξάνεται αντί να μειώνεται. Το να αυξήσουμε τους πόρους ε, δεν ε, θα αποτρέψει τη δολοφονία ενός ε, δημοσιογράφου που διεξάγει έρευνα όπως στη Μάλτα ή στην Τσεχία και δεν υπάρχει ακόμα καμία έρευνα παρότι το έχει ζητήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης Επίση υπάρχει στην Πολωνία συστηματική παρενόχληση των δικαστών. Θα μιλήσουν αρκετοί συνάδελφοι από αυτού. Αυτοί οι δικαστέ ε, αντιμετωπίζουν ε, μια συντονισμένη επίθεση ρητορική μίσου, προπαγάνδα ε, για να αποτρέψουν οποιαδήποτε ανεξαρτητοποίησή του. Ούτε καν ο επικεφαλής του Δικαστηρίου δεν είναι ασφαλή. Οποιαδήποτε περισσότερη πληροφορία μπορείτε να μα δώσετε για το θέμα αυτό θα ήταν εξαιρετικά ε, ωφέλιμο και πολύτιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Και τώρα η κυρία Ζίμπερ, Ζίμερτ. Uh, να ξεκινήσω με κάτι που ανέφερε ο Επίτροπος Τίμερμανς ε, στην παρέμβασή του. Θέλω όμως να το υπογραμμίσω και εγώ. Ο τίτλος της ανακοίνωσης του Ιουλίου είναι «Ενίσχυση του κράτους δικαίου». Γνωρίζουμε όλοι όμως, το είπατε κι εσείς, πως ε, αυτή η έννοια δίνει ίσω κάποιε ασφαλμένε εντυπώσει, διότι πολλοί λένε Α, ενίσχυση του κράτου δικαίου. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε βασίζεται σε νόμους. Αυτό όμως δεν αρκεί, διότι γνωρίζουμε και έχουμε βιώσει την εμπειρία αυτή σε τουλάχιστον δύο-τρει χώρε, ότι αν έχει την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μπορεί να συντάσσει νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αυτή τελικά να καταστρέφει τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών, άρα και τι κοινέ μα αξίε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε μια διαφορετική διατύπωση και να μην μιλάμε πλέον μόνο για κράτος δικαίου. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό ενδέχεται να παραπλανά κάποιες φορές. Επίσης, αυτό που είπε η Ρομπέρτα, θέλω και εγώ να το τονίσω, οτιδήποτε κάνουμε εμείς και ε, όποιες οδηγίες κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν, ε, η ρητορική μίσος ή τα προβλήματα για δικηγόρους, δικαστές και πολλούς άλλους ε, ε, από την κοινότητα των πολιτών δεν θα πάψουν να υπάρχουν προβλήματα και οι κυβερνήσει θα πρέπει να αντιδρούν σε αυτή τη ρητορική ε, και στην παραπληροφόρηση. Επομένως, πέραν των σαφών κανόνων, χρειάζεται και κάτι περισσότερο. Χρειάζεται μεγαλύτερος, περισσότερος διάλογος, ώστε με όλες τις διαφορετικές παραδόσεις να υπάρξει μεταξύ κρατών μελών συνεννόηση. Αλλιώς οι αξίες που έχουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, τι νόημα θα έχουν. Δεν είναι κάτι που έχουμε φεύρει εμείς. Όλες αυτές οι αρχές, οι αξίες προέρχονται από τα κράτη-μέλη και είναι κοινό αποδεκτέ. Επομένω, ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Ναι, πρέπει να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένε υποθέσει όπω αυτή τη Σλοβακία και Μάλτα. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση και να αποφύγουμε την ε, το ενδεχόμενο κάποιες μειονότητες να μην καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει κράτος δικαίου στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Κύριε για την ομάδα Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίαση του και για την κατάθεση αυτής της πρότασης. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μιλώ εκ μέρους ομάδας Renew κράτος δικαίου, δημοκρατία, θεμελιώδεις ελευθερίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι όμως και εισηγήτρια ε, για αυτή την πρόταση του DRF ε, και χαίρομαι που συζητούμε αυτή την πρόταση για έναν συνεκτικό μηχανισμό, διότι ναι με ένα πρόθυμα ε, το Συμβούλιο και αυτό, όπως και όλοι οι άλλοι, υιοθετούν την ίδια αυτή αντίληψη ότι πρέπει κάτι να γίνει. Να πω κάτι για τη διαδικασία καταρχάς. Θέλω να προειδοποιήσω ε, ότι θα είναι αρνητικό να υπάρξουν πολλαπλή μηχανισμοί. Θέλουμε ένα σύστημα μόνο με κοινά πρότυπα, όχι διαφορετικά για το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν. Άρα πρέπει να επεξεργαστούμε έναν ενιαίο μηχανισμό όπω είχε προταθεί και στην αρχή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Το λέμε κράτο δικαίου, λέγεται, αλλά πρέπει να καλυφθούν και άλλα στοιχεία. Μα αν καλυφθούν άλλα στοιχεία, α το πούμε. Α βάλουμε ε, τα ονόματα, ας κατονομάσουμε στο κείμενο ότι πρέπει να περιληφθεί το άρθρο 2 στο πλήρε πεδίο εφαρμογή. Το είπαν και συνάδελφοι. Ε, Εκστρατείε δυσφήμιση, ε, παρενόχληση δικαστών, κυνήγι μαγισσών ομοφοβικό. στην Πολωνία το είδαμε από το κυβερνών κόμμα. Η ακαδημαϊκή δημοκρατία στη... και το άσυλο κινδυνεύει στην Ουγγαρία, ε, όπου παρακάμπτεται το κοινοβούλιο, φήμωση και εκφοβισμός ε, των δημοσιογράφων. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Ρομπέρτα για τη μορισία ε, για έναν δολοφόνο και αυτό είναι πολύ σημαντική παραβίαση. Κύριε Βαντερλάιν λέει πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Μα δεν είναι εθνική ιδιαιτερότητα οι αξίε αυτέ. είναι ευρωπαϊκέ αξίε και είναι αδιαπραγματευτε. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά εθνικά συστήματα, οι αξίε μα όμω είναι κοινέ και πρέπει να τι προστηρίξουμε. Τέλο, η ομάδα μα ε, θέλει να συνεργαστεί μαζί σα Επίτροπε, προσβλέπουμε σε αυτό γιατί θέλουμε να είναι πρωταθλητής της δημοκρατίας του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους πράσινους η κυρία Τρίκ, η κυρία Ρένκε, συγγνώμη. Ναι, θα συνεχίζουμε έτσι να παίρνουμε τη σύγχυση, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε την ε, ε, ανακοίνωση. Νομίζω έγινε ήδη αναφορά στα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα. Χαιρόμαστε βεβαίω που προτείνει κάτι η Κομισιόν, αλλά όντω υπάρχουν μια σειρά από όπου το Κοινοβούλιο ήδη σε έκθεσή του ε, έχει πιο προχωρημένες θέσεις. Και για μας είναι σημαντικό ιδιαίτερα το θέμα του πεδίου είπατε ότι υπάρχει αυτό ο σύνδεσμό ο στενό, αλλά αν δείτε τι γίνεται παραδείγματο χάρη στην Πολωνία, όπου βλέπουμε ότι οι ακτιβιστές LGBTI ε, δέχονται επίθεση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί να μην είναι λοιπόν στο πεδίο αυτή τη ανακοίνωση, γιατί να μην καλυφθούν. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτού του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να του πούμε ότι αυτό αποτελεί μέρο του πεδίου των κράτου, του δικαίου των ευρωπαϊκών αξιών σε ό,τι αφορά του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε, είπατε ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε είναι ένα σημαντικό ε, θετικό στοιχείο στι εργασίε τη Κομισιόν. Γιατί να μην του δώσετε όμω και την ε, αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, για το monitoring, διότι αυτό είναι που θα δείξει ότι εδώ μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Δεν είναι απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν κατά των κρατών μελών. Υπερασπιζόμαστε ευρύτερα τι ευρωπαϊκέ αξίε. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι αυτό αυτή η στενή διασύνδεση με τον προπολογισμό της Ένωσης είναι κρίσιμη διότι μπορεί να, υπάρξει, να υπάρχουν διαδικασίες παραβάση αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα οδηγήσει σε ε, επιπτώσεις οικονομικές όταν ένα κράτος μέλος δεν σέβεται το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ευχαριστώ κύριο Σταρντίνο για την IND. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Άκουσα με προσοχή την ε, παρέμβασή σας. Μ' ακούτε? Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επιτροπή. Άκουσα με προσοχή την παρέμβασή σα και δεν μπορώ παρά να επισημάνω ένα σφάλμα ουσία από την πλευρά τη Επιτροπή. Μιλάτε για κράτο δικαίου, να θυμίσω ότι η βασική ευθύνη για την διαφύλαξη του κράτου δικαίου είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και των εθνικών του φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ω θεματοφύλακα των συνθηκών, έχει σημαντικό ρόλο να διαρματίσει υπ' αυτή την έννοια βέβαια, ε, και πρέπει να χρησιμοποιήσει τα διαδικαστικά συστήματα και τα νομικά μέτρα που προβλέπονται σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσει κάτω δικαίου, εφόσον το κάτω μέλο παραβιάσει τι υποχρεώσει του βάση του ευρωπαϊκού δικαίου. Όμω δεν συμβαίνει αυτό. Ούτε αυτό ακούσαμε σήμερα, ε, ούτε τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε τιμωρητική ή κατασταλτική στάση πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία να είναι εφικτά και να μπορούν να υλοποιηθούν τα κράτη-μέλη θα μπορούν ταυτόχρονα να είναι σε θέση να σέβονται τις συνθήκες. Βάσει της θητείας σας είδαμε πολλές διαδικασίες ε, του άρθρου 7 να εκκινώνται. Επίσης ε, σε κάποιο δημοψήφισμα είδαμε να ψηφίζει ένα σημαντικό το μέλος να αποχωρήσει από την Ένωση. Και ανακοινώθηκε ότι στόχος ήταν η απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, προκειμένου η Μεγάλη Βρετανία να μην χρειαστεί να αποχωρήσει. Τελικά δεν πετύχαμε το στόχο μας. Εδώ λοιπόν τα διδάγματα είναι απλά. Ε, και οι ερωτήσει μου επίση. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριφέρθηκε σωστά ως προς το σεβασμό του κράτους δικαίου και μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα επιτυχίας, όχι μόνο πολιτικής επιτυχίας, αλλά και σε πολιτών που επέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δράσεις της αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ερωτήματα στα Ολλανδικά όμως θα τα θέσω. Ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση κύριε Τίμερμανς. Όμως ο τίτλος ήδη δημιουργεί πρόβλημα για μας. Ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ένωση. Πρόκειται για αντίφαση. Η διαφύλαξη του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ευθύνη όλων των κρατών μελών. Το κράτος δικαίου έχει να κάνει με το δίκαιο της κάθε χώρας. Είναι κάτι που σχετίζεται λοιπόν με τα κράτη-μέλη και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μιλάτε για μέτρα όπως η ενίσχυση της κουλτούρας του κράτους δικαίου από την κοινωνία των πολιτών, τα μίντια, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τα συστήματα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως λέτε, πολύ σωστά, ότι πρέπει το κράτος δικαίου να προβλέπει πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρεμβαίνουμε όσο γίνεται λιγότερο από το εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, εσείς ε, ουσιαστικά δημιουργείται μια υπερστρουκτούρα την Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τα πάντα. Δεν βλέπετε δηλαδή εδώ παρέμβαση όταν παρεμβαίνετε εσεί. Ε, συμφωνείτε ότι τα προληπτικά αυτά μέτρα στα μέσα ενημέρωσης και στον τομέα της εκπαίδευσης επίσης ε, μοιάζουν ουσιαστικά με δόγματα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, μιλάτε για τη συμφωνία του Κράτου δικαίου, για, τη, την σημασία του κράτου δικαίου, λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο ε, κάποια κόμματα τα οποία αφισβητούν ή ε, επιλούν αυτές τις αξίες θα πρέπει να απαγορευτούν ή όχι. Μα ε, είναι βασική αρχή του κράτους δικαίου, κύριε Τίμερμαντς. Πρέπει να έχουμε μια υγιή ανταλλαγή απόψεων, ελεύθερη και όχι απαγορεύσεις. Μπορείτε δηλαδή να, να αποκλείσετε ευρωπαϊκά κόμματα, κόμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Ένστ και από την ΚΟΕ. Ε, Καταρχάς, ε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Κύριε Τίμερμαν, σας βλέπουμε με μεγάλη χαρά και Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη και κάποιες κυβερνήσεις που δεν σας συμπαθούν και τόσο πολύ ε, και αυτό κάποιες φορές έχει και πολύ αρνητικές επιπτώσεις, οφείλω να πω. Ε, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, είδαμε και ακούσαμε ότι ουσιαστικά είναι ένα είδος ε, ετερόκλητου προϊόντος που μπορεί κάποιος να βάλει κάτι, να βγάλει κάτι. Είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί ενίοτε. Αυτό το σύστημα, έτσι όπως το έχετε πλέξει, αυτό το χαλί με τα πολλά χρώματα, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να οδηγήσει σε μια εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά τα ποινικά ζητήματα και την αμοιβαία αναγνώριση. Εδώ το ζήτημα είναι ακαθόδες και δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Ε, παραδείγματο χάρη ε, δικαστήριο, κάτι το ε, αποφάσισε σε σχέση με την Πολωνία, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν για τι απελάσεις, τις εκδόσεις. Φαίνεται ότι τελικά δεν λειτουργεί το δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σωστό τρόπο. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές αξίε και αξιολογήσει σε ό,τι αφορά το δίκαιο. Λέμε ότι είμαστε μια κοινότητα και μένουμε όλα μόνο στα λόγια. Πώς μπορούμε όμως να σταθεροποιήσουμε αυτό το σύστημα, να υπάρχει παραδείγματο χάρη η αμοιβαία αναγνώριση ε, στον ποινικό τομέα, στο ποινικό δίκαιο. Και επίσης, ε, επειδή υπάρχει πάντα αυτό το δούνε και λαβίν, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό κυρώσεων στο εσωτερικό της Ένωση, θα ήθελα να ε, μου πείτε ε, τι δυνατότητες ε, προσφέρονται όταν υπάρχουν χρήματα. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα και αν είμαστε χαλαροί και άνετοι δεν μας ενδιαφέρει και τόσο η παραβία στροπέν δικαιωμάτων. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτού του μηχανισμού επιβολής κυρώσεων. Ακούσατε με πολύ ενδιαφέρον κύριε Τίμερμανς φαντάζομαι τις ερωτήσεις ε, ε, και σίγουρα είδατε ότι πολλοί εκφράζουν ε, την ικανοποίησή τους για το έργο σας γιατί το κρατός δικαίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά ψηφίσματα, έχετε δείξει στένο στον τομέα αυτό, το ξέρουμε. Τώρα όμως έχετε εσείς το λόγο για να απαντήσετε και επειδή με Είμαστε 30 υπόλοιποι που θέλουν το λόγο. Παρακαλώ να μας δευκολύνετε και εσείς σας απαντήσει. Ευχαριστούμε. Κάποια από τα ερωτήματα μάλιστα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, θεμελιώδη, μπαίνουν στον πυρήνα των ζητημάτων. Είναι κάπως ηρωνικό ότι δύο ομιλητέ εδώ που εκπροσωπούν κόμματα που λένε ότι είναι τα μόνα που εκπροσωπούν τη φωνή του λαού δεν δέχονται ένα ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο κράτο δικαίου. ...είτε πρέπει να είναι περιορισμένο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Ενώ το Ευρωπαρόμετρο δείχνει ότι 89% του πληθυσμού τη Ένωση θεωρεί ότι το κράτο δικαίου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κάτι με το οποίο πρέπει να εμπλέκεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το κράτο μέλο. Το κράτο μέλο, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ακούσετε λοιπόν το λαό, αυτή τη θέση πρέπει να εκπροσωπείτε. Και όχι να το κάνετε εθνικό ζήτημα. Τώρα βεβαίως υπάρχει το θέμα του γιατί. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει και να εμπλέκεται σε αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με την ουσία της Ένωσης ως ένα σχέδιο ειρήνης. Διότι εάν δεν έχουμε μια κοινή κατανόηση σε ό,τι αφορά το σεβασμό, των κανόνων, των νόμων, των συνθήκων, τότε θα ενεργοποιήσουμε και πάλι μια Ευρώπη κρατών αντίον κρατών, λαών αντίον λαών. Αυτό είναι το νόημα της ιδέας της Ένωσης. Να μην έχουμε πια αντιπαράθεση ε, και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι είναι όλοι δίκαιοι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Στον νόμο. Παλιά κρατημέλη, νέα κρατημέλη, μικρά κρατημέλη, μεγάλα κρατημέλη, ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό αυτών των χωρών. Εάν λοιπόν το ξεχάσουμε αυτό και πούμε α αφήσουμε τα κρατημέλη να αποφασίσουν πώ θα ερμηνεύσουν την, την νομοθεσία, α μπορούν οι κυβερνήσει να ελέγχουν του δικαστέ, τότε ε, η ουσία, η βάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πάβει να υπάρχει. Δεν μπορώ να το πω πιο σαφώ. Και βεβαίω είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι όταν δεν έχουμε ίση εφαρμογή, ίδια εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη, δημιουργούνται ανισότητε. Όταν έχουμε μια κοινή αγορά, κάθε επιχείρηση σε αυτή την κοινή αγορά πρέπει να μπορεί να βασίζεται στην ενιαία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ποιο ελέγχει την εφαρμογή αυτήν. Ο εθνικό δικαστή. Ο εθνικό δικαστή λοιπόν είναι ταυτόχρονα και Ευρωπαίος δικαστή όταν ένα δικαστή είναι ε, τον έλεγχο μια εθνική κυβέρνηση, δεν έχουμε πια την εγγύηση ότι θα εφαρμοστεί ενιαία η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρχίζει και η ε, εσωτερική αγορά να αποσυντίθεται. Είναι πολύ απλό αυτό, πολύ, πολύ σαφέ. Όπω η κυρία Ζήπελ όμω, δεν είναι μόνο θέμα νόμων. Το κράτο δικαίου, η ελεύθερη κοινωνία, η ανοιχτή κοινωνία, η δημοκρατία είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε μόνο σε νόμους. Έχει να κάνει με την πολιτική συμπεριφορά, την κοινωνική συμπεριφορά, τη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό τα ζητήματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να έχουμε κράτος δικαίου εάν δεν έχουμε ανεξάρτητο τύπο που να μπορεί να αναφέρει ανεξάρτητα το τι συμβαίνει και δεν μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητο τύπο αν δεν υπάρχει κάποιο δικαίωμα που να προστατεύει του δημοσιογράφου. Ο νόμο να του προστατεύει. Το ίδιο ισχύει και με την κοινωνία των πολιτών. Αν δεν έχουμε μια κοινωνία των πολιτών ε, ζωντανή, όπου εκφράζουν οι πολίτε τι απόψει του, ε, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρο λοιπόν τη προσέγγιση μα τα επόμενα χρόνια. Θέλω να είμαι σαφή. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά θεωρούν ότι η ανακοίνωση αυτή είναι να βγει προ σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Α γίνει αυτή η συζήτηση να τη συνεχίσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να συζητούμε μαζί στα επόμενα πέντε χρόνια. Όπου μπορούμε θα πάμε παραπέρα, θα βελτιώσουμε τα κείμενα. Διότι πραγματικά θυμάμαι, ε, πιστεύω, ότι ο ίδιος ο ιστός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βάση της, διακυβεύεται αν δεν μπορούμε να προθέσουμε το κράτος δικαίου, την προστασία της ελευθερίας του τύπου, της προστασίας της κοινωνίας των πολιτών, τη δημοκρατία, όλα αυτά συνδέονται. να πω και κάτι για το ρόλο των κρατών μελών. Τελικά, οι μόνοι που μπορούν να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου δια... προστατεύεται είναι οι πολίτες ε, των κρατών μελών. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο το επιθυμεί. Τελικά όμως η κατεύθυνση μιας χώρας καθορίζεται από τους πολίτες της. Έχουμε όμως και εμείς την ευθύνη να εξηγήσουμε στους πολίτε ποιε είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων που παίρνουν. Ένα παραδείγματο χάρη, η συμπεριφορά μιας κυβέρνησης οδηγεί σε μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα της στο περιθώριο της Ένωσης. Και φοβούμε ότι συχνά αυτό γίνεται χωρίς να το θέλουν αυτό οι πολίτες των χωρών αυτών. Και ο μόνος τρόπος για να είναι σαφές αυτό είναι μέσω της δημόσιας συζήτησης, μέσω των μίντια, της κοινωνίας των πολιτών. Συνδέεται λοιπόν και αυτό με τις προσπάθειες που κάνουμε για να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών. Ε, αυτό είναι προφανές. Θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση προφανώς και για την ελευθερία του τύπου πώς μπορούμε να μειώσουμε την πίεση ε, στον, πάνω στον τύπο, ε, να δούμε και επίσης και από οικονομικής πλευράς ε, πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί μόνο έτσι μπορεί να είναι ελεύθερα. Μπορεί να το δει αυτό το Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα χρόνια. Για άλλη μια φορά να πω ότι δεν είναι μόνο θέμα δικαίου και νόμων αλλά γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το δίκαιο. Είναι το μόνο μέσο που έχουμε για να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται οι συμπολίτε μα. Ο νόμο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο νόμο και ο σεβασμό του νόμου είναι η μόνη πραγματική ασπίδα που έχουμε για να προστατεύσουμε του πολίτε. Υπογράφοντα λοιπόν τι συνθήκε τη Ένωση, επικυρώνοντά τι δημοκρατικά, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται δεν μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιείτε το επιχείρημα της κυριαρχίας για να πείτε κυριαρχία σημαίνει ότι εγώ ε, ε, θα αποφασίσω εάν εφαρμόζω ή όχι ή πώς εφαρμόζω τις διεθνείς συμβάσεις που έχω υπογράψει. Η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων και αυτό το, αυτό το καθήκον το έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά. Νομίζω πως εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια έχω δείξει ότι το παίρνω πολύ σοβαρά, ανεξάρτητα από τις όποιε επιπτώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Τίμερμανς. Συνάδελφοι, ο μόνος τρόπος να προλάβουμε στα επόμενα 45 λεπτά είναι η κάθε μια και ο καθένας να περιοριστούν σε ένα λεπτό. Ακριβώς. Παρακαλώ, προσέχετε την ποσότητα των λεγόμενων σας. Περιορίστε το ε, πόσο θα μιλήσετε στο ένα λεπτό. Αφαιρέστε ότι ξεπερνάει το λεπτό. Θα προσπαθήσω να τηρήσω μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Πέσατε. Είστε καλά. Ο κύριος Ιππέγγι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από την Ουγγαρία. Ισφαν Ιππέγγι. Πολύ καλό να ενισχυθεί το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιέπαινη προσπάθεια. Όμω δεν έχω πολύ μεγάλε ελπίδε σε σχέση με τι εμπειρίε τη τελευταία διετία. Από την ανακοίνωση αυτό που μα λείπει είναι ένα σαφή ορισμό του τι εννοούμε. Δεν υπάρχει ένας αντικειμενικός ορισμός του κράτους δικαίου. Εάν δούμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό καθεστώς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε μια ποικιλία διαφορετικών νομικών συστημάτων, πολιτικών φορέων και όλα μπορούν να είναι δημοκρατικά. Αυτό που είδαμε είναι να γίνεται κατάχρηση του όρου κράτος δικαίου και μάλιστα κατά συγκεκριμένων κρατών μελών, ειδικά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Κατά την άποψή μου λοιπόν εδώ γίνεται κατάχρηση της έννοιας του όρου και καταστρέφει την ισορροπία του κράτους δικαίου. Εάν γίνει ιδεολογικό όπλο κατά μιας ιδεολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Μπούρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως τα ξέρετε, στην Πολωνία από που έρχομαι, ο κόσμος σας γνωρίζει ως είτε ως ε, τον ε, υπαριθμόν ένα εχθρό, είτε ως τον υπαριθμόν ένα προστά, προστάτη και εγγυητή των δικαιωμάτων μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την, ε, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρετε πώς, μπορείτε να, πώς θα μπορούσατε να πιθαναγκάσετε τις κυβερνήσεις για την κατανομή των ε, διαφορών κονδυλίων και για το σκάνδαλο Πιέβιακ, κάποια πράγματα που μας έχουν ανησυχήσει πολύ για το κάτω δικαίου στην Πολωνία. Ξέρω ότι ο εκπρόσωπό σα γνωρίζει το θέμα. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της Επιτροπής. Πολύ γρήγορα να σχολιάσω ότι ο ε, κ. Σκουεδιάκ είναι Υπουργό Δικαιοσύνη στην Πολωνία, υπεύθυνο για το δικαστικό κλάδο και καθερέθηκε αφού δημοσιεύτηκε μια ε, υποτιθέμενη συζήτησή του από το Facebook που μπορεί να αποτελεί μέρος εκστρατείας εκφοβισμού των δικαστικών λειτουργών με συντονισμό του το Υπουργείο Δικαιοσύνη το ίδιο. Ευχαριστούμε κύριε Κόρμπετ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σα. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση, ήδη το θίξατε μέρη, για τον προπολογισμό τη Ένωση. Είμαι εισηγητή τη ομάδα Renew για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Προπολογισμών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώ θα τα συνδυάσετε αυτά με την πρότασή σα τι δημοσιονομικές συνέπειες θα υπάρχουν και τι ε, μέτρα για την τήρηση του κράτους δικαίου. Ευχαριστούμε, κύριο Λαγκοντίνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει. Είπατε ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Να την συνεχίσουμε, αλλά η κυρία Φαντεν Λάιεν είπε ότι το κράτος δικαίου μας ενδιαφέρει πολύ. η Δεύτερη ερώτηση. Είπε ότι ποτέ δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις ε, στον τομέα αυτό. Τι εννοείται ακριβώς, ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις διάκρισης. Ε, ε, θεωρείτε ότι για το κράτος δικαίου γίνεται λόγος εδώ για διακριτική μεταχείριση σε βάρος κάποιας χώρας. Δεν θέλουμε εκπτώσεις στον τομέα της Προστασία του κράτου δικαίου, ούτε από εσάς την κυρία Φοντελάν και ε, για τα τεχνικά ζητήματα. Μιλήσατε για τη στήριξη τη κοινωνία των πολιτών διαμακρών. Συγκεκριμένα, ποια εργαλεία πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων έχουμε, ώστε παραδείγματο χάρη να στηρίξουμε ΜΚΟ στην Ουγγαρία όταν καταπιέζονται. Νομίζω ότι καλό είναι πλέον να πάρει την ευθύνη η ε, Κομισιόν και αυτή να ρυθμίσει τα πράγματα για τις ΜΚΟ. Ευχαριστούμε ο κύριος Βυσνιεύσκη. Η κυρία Βυσνιεύσκη. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, ε, σας άλλαξα φίλο. Δεν πειράζει. Panie e, Κύριε Επιτροπέ, καλά σας βλέπω. Ε, στη διάρκεια των θερινών διακοπών ε, περίμενα να πάρετε κάποια απόσταση από αυτά που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Αυτό έλπιζα τουλάχιστον. Λέτε από τη μια πλευρά ότι θα πρέπει στην Ένωση να ενισχυθεί το κράτος δικαίου. Ας δούμε. Ας δούμε, κύριε Επίτροπε, τι γίνεται στη χώρα σας, στην Ολλανδία. Εκεί υπάρχει το συνταγματικό δικαστήριο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς θέλετε λοιπόν να εναρμονίσετε, να παγιώσετε τους νομικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου, όταν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές ε, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Πέραψατε να σας πω ότι όταν ε, ήταν προηγούμενη κυβέρνηση στην εξουσία στην Πολωνία, εσείς ήσασταν ο πρώτος, στο πρώτο μέτωπο ε, της Αντίθεση ε, και δεν μπορούσατε καν να ακούσετε αυτά που λέγονταν ε, για τα χρήματα και το πώς αντιμετώπιζε η κυβέρνηση τη χώρα σαν να είναι εταιρεία της. Είναι 30 άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ένα λεπτό έχει ο καθένας. Ε, σας παρακαλώ. αν το έχετε γραπτό στο κείμενο τότε συντομεύστε το. Τι να σας πω. Η κυρία Πιόρκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα θέλω να πω. Κάποια τα είπαν και οι συντονιστέ άλλωστε. Πρώτα απ' όλα το πεδίο. Το κράτο δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία δεν συνδέονται μόνο μεταξύ του. Δεν συνδέονται απλά. Είναι, είναι αδιάρρηκτα. Ε, δεν μπορούν να διαχωριστούν. Γι' αυτό δεν αναφέρεται παρκώς έχουμε μιλήσει για την ομοφοβία, για την, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών, των προσφύγων. Ε, πολλές ελπίδες στην κοινωνία των πολιτών ε, δεν μπορούν να δράσουν δεν μπορούν να δράσει η κοινωνία των πολιτών σε κάποια κράτη-μελίδη. Θα πρέπει λοιπόν να τα συνδέσουμε αυτά, όχι απλά να τα συνδέσουμε, να καταλάβουμε ότι είναι ένα. Το είπαν και κάποιοι συντονιστέ. Θέλω να το υπογραμμίσω δεν επιλύεται αυτό στις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Και το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με την απάντηση. Πολύ αδύναμη η φρασιολογία. Να υποστηρίξουμε, να εξετάσουμε, να μελετήσουμε. Όχι. Πρέπει να τα συνδέσουμε αυτά και με τις τον προπολογισμό της Ένωσης και με τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάμοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα σας ευχαριστήσω και που παρουσιάσατε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ με φόβο βλέπω ότι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάχρηση εξουσίας στην Πολωνία. Δώσατε και παραδείγματα, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Όμως ε, το πιο πρόσφατα παράδειγμα είναι μια κατάσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας μου όπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Ισαγγελέας, ο Γενικός Ισαγγελέας ε, ε, έχουν, ε, είδαμε ότι είχαν ε, ένα ολόκληρο στρατό από τρόλ στο ίντερνετ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούν τωρική μίσος η ίδια κυβέρνηση στα μίντια. Είναι πραγματικά από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας ο, άντρα άντρας μου δολοφονήθηκε ε, λόγω αυτής της τρορικής μίσους φέτος τον Ιανουάριο. Η πολωνική κυβέρνηση ε, δεν εκτελεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεν τις σέβεται. Είναι πραγματικά το πιο επικίνδυνο ε, όπλο αυτή τη στιγμή στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Στα βουλγαρικά θα θέσω το ερώτημά μου. Πραγματικά, η ανακοίνωση από τις 17 Ιουλίου είναι εντυπωσιακή. Προτείνεται την πρόβλεψη ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη πώς θα συνδυάζεται αυτή η έκθεση, έκθεση με την συνεργασία και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και την τήρηση του κατούς δικαίου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπάρχουν ε, για τις δύο αυτές χώρες τα τελευταία 12 χρόνια και δεν δίνουν αποτέλεσμα. Μην πω ότι ήταν και αντιπαραγωγικοί οι μηχανισμοί αυτοί. Έγιναν δηλώσεις ότι κάτι καταφέραμε, αλλά όχι αυτά αποτελέσματα. Τι θα γίνει. Είναι ο μηχανισμός αποτελεσματικός. Ευχαριστούμε. Η κυρία... Παγάθα Ορτουντούα, ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερος για την πολύ σαφή ε, παρουσίαση που έβριθε πολύ ενδιαφερουσών ιδεών για την κυρία Ιντβέλτ. Ε, δύο πολύ σημαντικά θέματα τίθενται ότι μπορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στο κράτος δικαίου να καταστραφούν από τις ε, πολιτικές πλειοψηφίες όταν ε, παραδείγματος χάρη μια κυβέρνηση ή κάποιο κρατικό φορέα και παρακρατικό φορέα που όμως έχει κάποιες αρμοδιότητες και δεύτερον οι δικές μας αξίες, οι δημοκρατικές αξίες είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο η ελευθερία συνείδησης όταν απέναντι στον νόμο και πολλές άλλες αρχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες Επομένως, ε, ε, ή θα πρέπει ε, να έχουμε κράτος δικαίου που θα είναι ανελεύθερο ή θα βασίζεται σε συγκεκριμένη ταυτότητα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ισχύει. Γι' αυτό, κυρία Ινβέλ και κυρία Ζίπελ, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μηχανισμούς, γιατί αν δεν αξιοποιήσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ε, θα μπορούσαμε ουσιαστικά ε, το μόνο που έχουμε να είναι κάποια χαρτιά πίσω από τα οποία κρύβονται οι κακές πρακτικές αυτών που ε, ουσιαστικά προσπαθούν να παραβιάζονται τα αδιαπραγμάτευτες αυτές αξίες και πρέπει να συνεχίσετε αταλάντευτα το έργο σας κύριε Τίμερμανς, κύριος Τσάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχετε κατηγορήσει επανειλημμένως στην Πολωνία λέγοντας ότι η διαδικασία διορισμού δικαστικών λειτουργών είναι πολιτικός ε, υποκινούμενη. Όμως, αυτή τη στιγμή, τους δικαστικούς λειτουργούς ε, τους ορίζει ένα συμβούλιο το οποίο αποτελείται από λειτουργούς. Ε, επί παραδείγματι σε άλλε χώρε, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία. Όχι απλώ οι πολιτικοί απευθεία διορίζουν του δικαστικού λειτουργού, αλλά έγιναν οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί. Όπω στη Γερμανία. Στην Αυστρία διορίζονται από τον πρόεδρο βάσει προτάσεων τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Πού είναι ακριβώ ε, η συμμεταχείριση, κύριε Πρόεδρε. Εδώ φαίνεται ότι δικαστικό, ε, ο δικαστικό κλάδο στην Πολωνία είναι λιγότερο επηρεαζόμενο από την κυβέρνηση και τα πολιτικά από τις άλλες χώρες. Κι όμως εσείς συνεχίζετε να παρουσιάζετε ε, επιχειρήματα λαϊκιστικά κατά της Πολωνίας. Εδώ λοιπόν, τι έχετε να πείτε για ένα πολιτικό σύστημα όπου πολιτικοί απευθείας διορίζουν δικαστικούς και πώς το συγκρίνεται με το πολιτικό σύστημα, όπου οι δικαστές διορίζουν δικαστές. Και έπειτα είπατε πάρα πολλά, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, διαβάζετε. Ε, δεν μπορείτε να διαβάσετε όλο σας το κείμενο. Έπρεπε να το ξαναδιαβάσετε αλλιώ για να προλάβετε σε ένα λεπτό. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Μπορείτε να πείτε, Πρόεδρε, τι κάνετε για να προσπιστείτε τους πολίτες τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία όταν προσπαθούν να δηλώσουν και τα δικαιώματά τους. ακούς το που παίζει ε, το Κομισιόν για την προστασία πρόσπιση του Κράτου δικαίου. Η ελευθερία των πολιτών ε, δεν κάνει κάτι η Ευρώπη γι' αυτό. Μέρες φορές υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν, δεν δέχεται να, αποφασί, να, να εφαρμόσει απόφαση δικαστηρίου. Αυτό διακυβεύει την ασφάλεια των πολιτών. Δεν αισθάνονται ασφαλεί. Εμεί έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, να, να προσπίσουμε την ασφάλειά του. Όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχουν μέλη του Υπουργείου Δικαιοσύνη που είναι εμπλεγμένα σε ένα δίκτυο ρητορική μίσου στο διαδίκτυο, είμαστε υπεύθυνοι εμεί για να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα είναι ασφαλεί. Ε, ότι οι πολίτε θα είναι ασφαλεί, μάλλον. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρί κράτο δικαίου. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η κυρία Σάντος. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Θα χρειαστείτε τα ακουστικά σας. Καταρχάς να χαιρετήσω την ε, τόλμη σας και τις ε, αποφασιστικές κινήσεις για την προστασία του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου χωρίς ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Σε αυτό συμφωνούμε πιστεύω όλοι. Το να προστατεύουμε την κοινωνία των πολιτών, το να προστατεύουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους ακτιβιστές στην πράξη είναι θεμελιώδους σημασίας. Όμως δεν έχουμε κονδύλια. Δεν έχουμε αρκετά από τον ετήσιο προπολογισμό. Χρειάζονται περισσότερα. Χρειάζεται τη στιγμή που δέχονται πιέσεις, τη στιγμή που είναι θύματα ε, καταναγκασμού και, και άσκησης πιέσεων, τότε να υπάρξει σαφής αντίδραση, ξεκάθαρη αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω λοιπόν να, σας, να μας πείτε. Τι προβλέπετε για την κατάρτιση μελλοντικών δράσεων, για την προστασία αυτών των ακτιβιστών που δέχονται πιέσεις, καταπιέζονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως εδώ στην Ήπειρο αυτή όπου εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη δράση σας, για την προστασία της χώρας μου, της Ρουμανίας. Ε, και που σταθήκατε στο πλευρό της κυβέρνησή μα, όποτε χρειάστηκε. Ξέρουμε ότι όλοι έχουν τεράστιες προσδοκίες για την επίτευξη αποτελέσματο. Αυτό το νέο πολιτικό κύμα και είμαι μέλος από ένα πολύ ε, νέο κόμμα, ε, το νέο μας λοιπόν κόμμα και ο συνασπισμό μας θέλει να γνωρίζει πώς μπορούμε να προσπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά το μηχανισμό. Θέλουμε κριτήρια τελείως σαφή. Αυτά. Μιλάω για την κοινωνία των πολιτών. Έχουν δώσει μάχες μαζί με τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην όλη προσπάθεια αξιολόγησης. Και επιτά πότε αναμένεται ο μηχανισμός να λειτουργεί πλήρω, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και των αποτελεσμάτων μας. Ευχαριστούμε κύριε Φέστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνσα. Μιλήσατε για το κράτος δικαίου και την κοινωνία των πολιτών που δέχεται επιθέσεις και πράγματι το είδαμε στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, που εντάξει υπήρχαν και κάποιοι βίαιοι διαδηλωτέ μεταξύ αυτών, αλλά ήταν και πολλοί περισσότεροι ειρηνικοί διαδηλωτέ οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση. Ε, και επομένως πότε θα ξεκινήσετε την ε, σχετική διαδικασία κατά της Γαλλίας ε, γιατί είναι επίθεση αυτό που συμβαίνει κατά της των πολιτών στη Γαλλία. Επίσης με βάση της αρμόδιας γερμανικής υπηρεσίας έχουμε αύξηση της εγκληματικότητας και ιδίως στον τομέα της βίας σε βάρος γυναικών και μάλιστα δυσανάλογα υφίστανται βία γυναίκες μετανάστρες. Η ερώτησή μου είναι αν μπορείτε να εξασφαλίσετε προστασία ε, και προστασία ιδίως για τις γυναίκες στη Γερμανία για να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στρίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε περισσότερου και καλύτερου τρόπου για την προστασία του κράτου δικαίου στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και αποτελεσματικότερε διαδικασίε βάσει του άρθρου 7. Στην τελευταία θητεία, το Κοινοβούλιο τήρησε μια θέση πολύ αποφασιστική βάσει τη έκθεση Αρχεντίνη και ζήτησε από, την, από το Συμβούλιο να εκκινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7. Όμω, τώρα περιμένουμε την ε, συνέχεια και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη επιφυλάσσονται, ε, ανταλλάσσουν επικριτικά σχόλια αντί να κάνουν κάτι για το κράτο δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, δεν μπορεί να λάβει περισσότερο χειροπιαστή δράση για να το, πάρει το ρόλο του το Συμβούλιο λίγο πιο πολύ στα σοβαρά. Δεν πρέπει ε, να λάβετε υπόψη και την τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου για τις διαδικασίες του άρθρου 7 ε, έτσι ώστε να περάσει λίγο και η δική μας άποψη στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαβάρμα, ο οποίο είναι Γενικό Συγγετής για το θέμα γενικού του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Τίμερμαντς, η βάση για τη συζήτησή μας θα μπορούσε να είναι εξή. Πρέπει να έχουμε έναν σφαιρικό μηχανισμό ή κάποια εργαλεία που θα πρέπει να εφαρμόζονται αναπερίπτωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα άθρα 2 και 7 της συνθήκης δεν εφαρμόζονται διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις ή κυρώσεις εκτός αν υπάρχει ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Και βεβαίω δεν πρόκειται να αλλάξει η κυρωσει εκτο αν υπαρχει ομοφωνια ολων των κρατων μελων και βεβαιω δεν προκειται να αλλαξει η συνθηκη Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το συνδέσουμε με τα χρήματα. Και ο προπολογισμό είναι ο μόνο τρόπο για να γίνει αυτό. Όμω, ο προτινόμενο κανονισμό ε, σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου και τι παρατυπίε και τι ελλείψει είναι αποτελεί μέρο του πακέτου πραγματεύσεων στο MFF, στο το πολιτισμό πλαίσιο. Δηλαδή, είναι μια ομοιρία ε, διότι και πάλι χρειάζεται ομοφωνία εκεί. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν γι' αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ε, πρέπει πραγματικά να μπορέσει να λειτουργήσει. Ε, εγώ θέλω να λειτουργήσω. Ο κ. Γκλουξμάν έχει το λόγο, παρακαλώ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ κύριε, Αντιπρόεδρε. Είπατε το τη λέξη ότι πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις. επιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να κάνει την επιλογή μιας δημοκρατίας χωρίς ελευθερίας, όπω το Φίντε στην Ουγγαρία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν επιπτώσει και οι επιπτώσει πρέπει να είναι σαφεί. Όμω, αυτή τη στιγμή το κλίμα στην Ουγγρική και στην πολιτική κυβέρνηση είναι ότι οι επιπτώσει δεν υπάρχουν. Τελικά αυτοί αποφασίζουν ε, σε ό,τι αφορά το πακέτο που συζητείται μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η εντύπωση ατιμορρησία, δημοσιονομικά, ποιε θα είναι οι επιπτώσει για την παραβίαση του κράτου δικαίου. Για να το πω έτσι απλά και ευθέω. Μπορεί κάποιος ε, να αρνηθεί τι αρχέ τη Ένωση θα πρέπει όμως τότε να απαρνηθεί ε, και τα κονδύλια και τότε ίσως να σκεφτούν αλλιώ αυτές οι χώρες. Ευχαριστώ ο Σμέκα. Μέκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο που είναι εδώ σήμερα. Όπως πολύ σωστά είπατε, πολλοί από εμά νιώθουμε ότι το κείμενο τη Κομισιόν είναι να προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ότι δεν αρκεί αυτό, δεν πάει αρκετά μακριά για την προάσπιση των αξιών μας. Κάποιες από τις βασικές αδυναμίες αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Ε, δεν αρκεί δηλαδή κανείς να εποπτεύει ε, τα θεσμικά όργανα ε, και τη δικαιοσύνη, διότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, πολύ πιο ε, δευτερεύοντες, περιορίζοντας και των πολιτών, απειλώντας τους δημοσιογράφους. Δεν αρκεί λοιπόν ο νόμος. Προστατεύοντας το κράτο δικαίου το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπής θα προστατεύει αυτόματα και την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν φαίνεται όμω αυτό στο κείμενο, δεν κατοπτρίζεται. Δεν είναι βέβαια το πώ θα το αναφέρουμε, αν θα μιλήσουμε για δημοκρατικά και δικαιώματα, δικαιώματα στο κείμενο, να το πούμε στο κείμενο. Ποια είναι τα μέσα που έχουμε για να τα εξασφαλίσουμε αυτά. Τα συγκεκριμένα, αν μπορείτε να μα πείτε κάτι από αυτού, θα ήταν πολύ καλό. Η κυρία Κένκο έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη θέση που αναλάβατε. Θα ήθελα να μιλήσω για τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, Συνήθω γι' αυτό μιλάω, δηλαδή, αλλά σήμερα θα μιλήσω για κάτι άλλο. Το κράτο δικαίου μιλάμε πολύ γι' αυτό στο Κοινοβούλιο και πολύ σωστά, διότι είμαστε μια ένωση δικαίου, κανόνων. Ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστά να γίνουν σεβαστοί αυτοί οι νόμοι, όμως συχνά διαφωνώ με κάποιους από τους συναδέλφους για το πώς θα συμβεί αυτό, πώς θα παρέμβουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ε, η οποία δεν θα ποινικοποιεί τα κράτη-μέλη για πολιτικούς λόγους. Ε, και βέβαια υπάρχει και το θέμα της μετανάστευσης. Ζητούμε η κατανομή αρμοδιοτήτων εδώ να γίνει σεβαστή για αρμοδιότητε του καθενό δηλαδή. Μπορεί το Κοινοβούλιο να εξετάσει κάποια θέματα, αλλά οι κυβερνήσει είναι αυτέ οι οποίε έχουν τον πρώτο λόγο. Επιπλέον, χρειάζονται πολύ συγκεκριμένε ε, δράσει για να προστατεύσουμε τι αξίε μα παντού. Ε, στη Σλοβακία, στη Μάλτα, στην Πολωνία. Ε, εκεί βεβαίως είναι εύκολη στόχη αυτή. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ παρά να θυμίσω στα μέλη τη ΕΣΥΑΡ ότι πρέπει να σεβαστούν το όριο ομιλία ε, όπω όλοι οι υπόλοιποι. Σα είπα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, αν θέλετε να διαβάσετε, επαναδιατυπώστε το. Διαβάστε προηγουμένω το χαρτί σα πριν αρχίσετε να κάνετε ανάγνωση. Τι θα γίνει. Finish it, finish it. Ολοκληρώστε το. Έχετε ξεπεράσει κατά 45 λεπτά δευτερόλεπτα το χρόνο σα. Είναι κυρία, πρόεδρε. Ναι, κάνω τη δουλειά μου όμως. Ε, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε και την ΕΑΣΟ αμέσως μετά. Και μετά έχουμε την Ιουλίσα και τους διευθυντές της Ιουλίσσα και περιμένουν. Ολοκληρώστε. Ναι, ακούστε, όπως και στην Ισπανία με το θέμα της Καταλωνίας, ε, δεν πρέπει να συνεχίσει. Εκεί βλέπουμε ότι η Ισπανία δεν έχει επιπτώσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μία από τις λύσεις για να ενισχυθεί το ε, εργαλειοθήκη για, το κράτος δικαίου είναι η συνεργασία και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 2007 υπήρξε ένα μνημόνιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι μια πολύ καλή βάση συνεργασίας. Επίσης με τον καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε μέρος ε, ε διεθνών συμφωνιών. Υπάρχουν και άλλες ε, σημαντικές συμβάσεις για την παρακολούθηση των χωρών, ε, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Όμως ε, ε, στην σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων εκεί δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Θα υπάρξει η διεύρυνση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στι του συμβάσεις. Ευχαριστώ κυρία Ζίντσερ, ευχαριστώ πολύ λέει κυρία Ίντσιρ. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να χειροκροτήσω την προσπάθεια που έχετε κάνει για να υπερασπιστείτε τη, τα θεμελιώδη, τη θεμελιώδεις αξία μας εδώ. Ε, όμως ε, ε, δυστυχώς η δημοκρατία αυτή τη στιγμή αποσυντήθεται. Είδαμε την έκθεση ε, πέρσι που μας είπε ότι έχουμε πλέον και δημοκρατίες μη ελεύθερες όπως στην Ουγγαρία. Υπάρχουν σχετικές εκθέσεις. Τώρα, στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τον Ιούλιο μας υποσχεθήκατε ότι θα εξεταστεί ως το τέλος του 2020 το κατά πόσο η, ο αντίκτυπος των προβλημάτων στην εφαρμογή του κράτους δικαίου ε, απαιτεί ένα νέο μηχανισμό πέρα από τους υπάρχοντες κανονισμούς για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε για τι είδους μηχανισμό μιλάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χουκ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τίμερμανς, χιλιάδες πολίτε στη χώρα μου, την Ηνωμένο Βασίλειο, βγήκαν στου δρόμου για να προσπιστούν το κράτο δικαίου. Συμφωνείτε ότι αν προσπαθεί μια κυβέρνηση μια χώρα να καταστήλει το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του για ένα μήνα, δεν υπάρχει κανένα κράτο δικαίου και λειτουργία του. Ευχαριστούμε, κυρία Ντόνεφ. Ευχαριστώ, κύριε Τίμερμαντ. Είπατε και συμφωνώ απολύτω μαζί σα ότι το να προβλέπουμε νόμου δεν αρκεί για την ενίσχυση του κράτου δικαίου χωρί δημόσιο διάλογο και κοινωνία των πολιτών εύρωστη. Τι θα κάνετε εάν δεν υπάρχει πολιτικό διάλογο χωρί πολυφωνία μέσω μαζική ενημέρωση και χώρο για το δημόσιο αυτό διάλογο ή αν αποδυναμώνεται η κοινωνία των πολιτών όπω στην Ουγγαρία, τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση, διότι αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την κοινωνία των πολιτών. Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο λιανό τι εννοείται ακριβώς άμεση χρηματοδότηση. Και επίσης θα ήθελα να εξηγήσετε λίγο την ετήσια έκθεση για το κάτω δικαίου. Ε, πώς εννοείται την άμεση σύνδεση εδώ με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια για τη δράση σα για το κάτω δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην προηγούμενη και την μελλοντική σα θέση. Ε, είπατε για περισσότερη συνεργασία με την Επιτροπή τη βενετία. Να θυμίσω και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όμω, στο Στρασβούργο. Μπορείτε λίγο να πείτε περισσότερα για τη συνεργασία αυτή. Έχετε τίποτα νέε πρωτοβουλίε υπόψη. Ευχαριστώ. And, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Κέμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για ισότητα, μιλάμε για ίσες ευκαιρίες. Ε, ε, η, ισότητα δεν αντικατοπτρίζεται με τον τρόπο με τον οποίο απευθυνθήκατε σε δύο κυρίες προηγουμένως. Μισό λεπτό, λέει αλλά κάποιο πρόβλημα έχουμε με την διαμηνία. Εγώ σας άκουγα από τα ισπανικά, αλλά μάλλον κάτι άλλο ε, έγινε γιατί δεν είχαμε μετάφραση όλες τις επίσημες γλώσσες. Μπορώ να συνεχίσω δηλαδή. Μάλιστα. Τα ξαναλέω λοιπόν. Απευθύνθηκα σε εσά καταρχάς ε, να σας πω ε, την κυρία την κυρία Βυσνιεύσκα, ε, να τις μιλάτε καλύτερα, να τις ε, σέβεστε, γιατί μιλάμε για ισότητα ε, των δύο φίλων. Λοιπόν, μιλήσατε κυρίως, κύριε Τίμερος, για την Πολωνία, την Ουγγαρία και άλλες ε, πρώην κομμουνιστικές χώρες. Είναι ένα σύστημα δικαιοσύνη που δεν έτυχε πλήρους αναθεώρησης ίσως μετά από την ανεξαρτησία αυτών των χωρών. Εμείς, ξέρετε, νομίζω ότι μπορούμε να επιβιώσουμε καλύτερα στο μέλλον. Τι κάνατε εσείς όταν ε, υπήρχαν επιθέσεις κατά των κίτρινων γυλαίκων, γιατί δεν εφαρμόσατε το άρθρο τα κατά της Γαλλίας. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε ε, στις συναντήσεις που έχετε με εκπροσώπους από το Open Society, θεωρείτε πως ε, όλοι γίνονται σεβαστοί μόνο μία οργάνωση, η οποία από ό,τι φαίνεται πάει στρέφεται σε βάρος, κατά της ε, Πολωνίας. Κοιτάξτε, ε, δεν σέβονται κάποιοι συνάδελφοι τους κανόνες του παιχνιδιού, που τους σεβάστηκαν όλοι οι άλλοι. Και γι' αυτό, ως πρόεδρος είχα το καθήκον να διακόψω με όλο το σεβασμό προς τους νέους συναδέλφους και τον καθένα συνάδελφο, παρακαλώ και εσείς να δείξετε σεβασμό σε μας και να τηρήσετε τους κανόνες όπως τους τήρησαν όλοι οι άλλοι. Κάθε ένας από τους συντηρητικούς μίλησε διπλάσιο χρόνο από αυτόν και στη διάθεσή του. Ο καθένας από εσά τους συντηρητικούς το έκανε. Προσπαθήστε να ε, συγκροτήσετε το λόγο σας ή περικόψετε τον ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνετε, αλλά να σεβαστείτε και εσείς τους κανόνες. Αυτός είναι ο δικός μου ρόλος και το χρέος με εδώ. Να φροντίζω για την συμμόρφωση όλων προς τους κανόνες. Και έχουμε στην ίδια διάταξη δύο σημαντικά σημεία πριν ολοκληρωθεί αυτό το σημείο που φυσικά είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ λοιπόν να σέβεστε όλους, να σέβεστε και τον πρόεδρο όπως σας σεβόμαστε και εμείς. Μιλούν ταυτόχρονα πολύ. Ναι, μπορείτε να τα λέτε, αλλά με καλούς τρόπους. Ε, ναι, συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί μου φωνάξατε και με πληγώσατε. Πράγματι, με πλήγωσε το γεγονός ότι μου μιλήσατε τόσο με, με φωνές. ο Τζάκ, εμείς το μόνο που ζητούμε είναι τα τα Θα έχετε το λόγο. Λέω πρόεδρος, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο των μιλητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι πολύ σημαντικό που είπατε στη δεύτερη παρέμβασή σας, ότι τελικώς οι πολίτες είναι οι καλύτεροι προασπιστές του κάτους δικαίου. Εγώ έρχομαι από ένα κάτω ε, τη Ρουμανία που έχουμε πολεμήσει σκληρά για τα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Όμως, για να γίνει αυτό, Χρειάζεται ενημέρωση από ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολυφωνία αυτό. Τι θα κάνουμε για την ελευθερία για την πολυφωνία και πώς θα μπορεί ε, ο μηχανισμός για το κάτω δικαίου να βοηθά τους δημοσιογράφους να αντιμετωπίζουν την παραπολιοφόρηση, όχι μόνο εν ώψη εκλογών αλλά γενικότερα να προστατεύουν τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Κυρία Βόλαφ. μακρά η συζήτηση για ένα πολύ βασικό ζήτημα. Μία πτυχή θέλω να υπογραμμίσω. Σίγουρα είναι πολύπλοκη αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ απλό, ότι από το λαό ξεκινά το δίκαιο, αλλά το κράτος δικαίου ξεκινά από τις κυβερνήσεις. Άρα η αφετηρία μας είναι ο λαός ουσιαστικά και εκεί πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση για να καταλάβουν οι πολίτες μας ε, ποια είναι τα κόμματα και ποιες είναι οι συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο το κράτος ε, δικαίου. Και νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και καθόλου πολύπλοκα. Να μην υπάρχει αυτή η υπερβολική επιβάρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έπειτα μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω. Okay, thank you We have completed. This is our duty too. Try to make the best. Ωραία ολοκληρώσαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι, διότι αλλιώς ο μόνος τρόπος είναι κάποια στιγμή να σταματάμε και κάποιοι να μην μιλήσουν καθόλου και να μην μπορέσουν να ακουστούν, ενώ είναι δικαίωμά του. Λοιπόν, είχαμε πάνω από 30 άτομα που μιλήσανε. Μάλιστα, υπάρχει ακόμα κάποιος. Συγγνώμη. Τελευταίο λεπτό. Παρακαλώ, να είστε σύντομος. Θα μιλήσω στα βουλγαρικά. Ε, κύριε Τίμερμαντς, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει να κάνει με την πρόοδο που σημειώνεται για τις, ε, στις, πιο, στις λιγότερο ενεπτυγμένες χώρες, στις πιο αδύναμες. Είμαστε σε μια κατάσταση όμως η οποία αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται συνεχώς. Λέτε ότι η ελευθερία του τύπου δεν είναι εφικτή χωρίς κράτος δικαίου. Η διαφθορά υψηλού επίπεδου και οι παραβιάσεις είναι κάτι το οποίο διαπιστών, έχει διαπιστώσει τη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Υπάρχει ένα αυταρχικό καθεστώς, μια αυταρχική κυβέρνηση που αγνοεί ε, τις συστάσεις της ε, συνθήκη της, της ε, Επιτροπής της Βενετίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι, η, η, Εθνική Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη και τελικά είναι υποταγμένη στην εκκληστική εξουσία. Ε, τι θα κάνετε γι' αυτό, κύριε Τίμερμαντς. Κύριε Αντιπρόεδρε, το ερώτημά μου είναι ε, το εξή. Από το 2004 και μετά είμαι ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια μπήκα στην πολιτική ω ε, ευρωβουλευτή Ρωμά. Πρέπει να σα πω ότι για το ό,τι αφορά το μηχανισμό κράτου δικαίου, τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει τεράστια ανάγκη ε, και είναι πολλά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα για να μην φτάσουμε στη στιγμή που χρειαζόμαστε τέτοιο μηχανισμό. Έχω κάνει έρευνα 25 χρόνια στον τομέα αυτό ω ανθρωπολόγο, Πρέπει να είναι να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Ε, η υπηρεσία των θεμελιών δικαιωμάτων είναι ένα πολύ καλό ε, φόρουμ για να διαβαστούν οι εκθέσεις της ε, νέο μηχανισμό με νέα χρήματα Ω ακτιβίστη πέντε δικαιωμάτων πρέπει να σα πω ότι αυτό το εργαλείο δεν το, δεν θα το χρειαζόμασταν εάν δεν υπήρχε ε, δεν υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά από την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως πολιτικός σύντονος πρέπει να σας πω ότι έχετε ήδη πολλά εργαλεία στη διαθεσή σας που μπορεί να επιλύσουν τα προβλήματα για τα οποία συζητούμε εδώ σήμερα. Να το συνδέσουμε με χρήματα πάντως δεν είναι καλή ιδέα και πραγματικά πιστεύω ότι το, η στρατηγική για τους Ρώμα, ο φάκελος για τους ε, ε, το φάκελο Στοκχόλμης ε, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι περισσότερο από αυτού. Εάν ε, είχατε ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Είχαμε πολλές ερωτήσεις, ένα μεγάλο μακρύ γύρο ερωτήσεων και βεβαίως εντάξει η συζήτηση είναι και έντονη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τίμερμανς. Έχει λίγο χρόνο βέβαια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ που μου λέτε ότι με βλέπετε σε φόρμα. Ε, ξέρεις, σε αυτή την ηλικία όλα τα κομπλιμέντα είναι καλοδεχούμενα. Το είπατε όμως με φόβο στη φωνή σας. Ε, μην ανησυχείτε, θα παραμείνω σε φόρμα και δεσμεύομαι για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, παραμένω δεσμευμένος και βεβαίω την περιπράσπιση του κράτους δικαίου. Αποδείχθηκε ότι όσοι επικρίνονται ε, για παραβίαση κράτους δικαίου, αντί να απαντήσουν στις ε, κριτικές αυτές, δαχτυλοδείχνουν άλλους, διότι δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Γνωρίζουν ότι η κριτική αυτή είναι απολύτως αιτιολογημένη ένα από τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Ιντεβελτ αλλά και άλλοι εδώ και χρόνια και που θα, θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση σε, αυτό, ε, σε αυτήν την τακτική του να δαχτυλοδείχνουμε άλλου, θα ήταν το κάθε κράτο μέλο να βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Και αυτό είναι και το νόημα τη πρόταση αυτή τη ανακοίνωση. Είναι ο πυρήνα τη. Και αυτό θα βάλει τέλο στο να δαχτυλοδείχνουμε άλλου όταν κάποιο ε, κατηγορείται για κάτι. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα ε, να δεχθούν μια παρακολούθηση, μια έρευνα όταν μιλάμε για ζητήματα κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα συγκρίνουμε συχνά ασύγκριτα πράγματα μεταξύ τους. Λέμε ότι μια χώρα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, οπότε αφού επιτίθεται στο δικό μας συνταγματικό δικαστήριο ε, δεν μπορείτε να το κάνετε ή αιτιολογείται εμεί να, το, επιτεθούμε σε αυτό, εσεί δεν έχετε καν συνταγματικό δικαστήριο. Δεν λέγεται πουθενά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο, στη συνθήκη τη Ένωση ότι πρέπει να υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Όμω, τι λέει η συνθήκη, ότι τα δικαστήρια πρέπει να είναι ανεξάρτητα και πρέπει να υπάρχει ε, διάκριση εξουσιών. Και η Πολωνία αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να βάλει τα δικαστήρια υπό τον έλεγχο των κυβερνήσεων. Και να προσθέσω Τώρα μιλάω εγώ, εσείς μιλήσατε, μιλήσατε αρκετά. Δεν έχετε τον λόγο. Να προσθέσω κάτι. Οι Πολωνοί δικαστές επιτέθηκαν, δέχτηκαν επίθεση, καμπάνιες ε, συκοφάντησης. Γιατί, γιατί ήρθαν στις Βρυξέλλες και μου μίλησαν. Αυτό στα μάτια της κυβέρνησης είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται να μιλήσει ένα δικαστή σε ένα μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού έχουμε φτάσει τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένας δικαστής φοβάται να αποτελέσει αντικείμενο εκστρατείας μίσους μόνο και μόνο επειδή μίλησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, πριν από κάποια χρόνια θα ήταν ε, κάτι το οποίο θα μπορούσα καν να φανταστώ. Θα πρέπει λοιπόν να παίρνει σε τέτοιου είδου καταχρήσει εμεί να ορθώσουμε το ανάστημά μα. Και κάτι άλλο, διότι έγινε λόγο και το άρθρο 2. Η απόφαση του δικαστηρίου του Ιουνίου στην πραγματικότητα τι λέει. Το ότι το άρθρο 2 εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη-μέλη. Η ανεξαρτησία λοιπόν της δικαιοσύνης είναι κάτι που μπορεί να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους να κάνει ό,τι θέλει με το δικαστικό του σύστημα. Υπάρχει υποχρέωση στα πλαίσια της συνθήκης να γίνει σεβαστή η ανεξαρτησία των, της δικαιοσύνης. Και όταν προσπαθούμε να την νοθεύσουμε αλλάζοντας το, το όριο ηλικίας των δικαστών, τότε υπάρχει παρέμβαση. Και το λέει το δικαστήριο. Είναι ένα μήνυμα αυτό για όλα τα κρατημέλη όταν αυτά προσπαθούν ε, να νοθεύσουν την εξαρτησία τη δικαιοσύνη. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, για την ενιαία εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, διότι τα δικαστήρια εξετάζουν το πώς οργανώνονται οι εκλογές, πώς αξιολογούν τα, αξιολογούν τα αποτελέσματα των εκλογών λοιπά Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι στην καρδιά των δημοκρατικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει... Α, ναι, και για άλλη μια φορά να πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναλέμε. Όλο αυτό το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασίζεται σε τρία στοιχεία. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ένα απέναντι στο άλλο. Δεν μπορούμε να, λέμε, να μιλάμε για δημοκρατία, να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία και έχουμε πλειοψηφία εμεί και μπορούμε να παρακάψουμε το κράτο δικαίου ή να παραβιάσουμε θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό το επιχείρημα είναι απαράδεκτο. Είναι επιχείρημα που έχουν χρησιμοποιήσει δικτάτορε, δεκαετία του 30 στην Ευρώπη. Θέλω να σα θυμίσω ότι όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων υπό τον ναζισμό βασιζόταν στο δίκαιο, σε νόμους, αλλά ήταν ε, αντίθετο στα θεμελιώδη δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, αλλά βασιζόταν σε κάποιο νόμο. Έχουμε μια επιλογή, είτε θα έχουμε κράτος δικαίου, είτε θα έχουμε το, το να κυβερνάει κανείς με νόμους. Ξέρω βεβαίως ότι εδώ τώρα ίσως να ε, ενθουσιάζομαι υπερβολικά στη, στην παρέμβασή μου, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη μάχη που θα δοθεί τα επόμενα χρόνια. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας εδώ ε, να το αγνοούμε το θέμα. Ε, καλύτερο είναι να έχουμε καλές σχέσεις με όλους, με όλα τα κράτη-μέλη ε, ή να το παραβλέπουμε. Όποιες και είναι επιπτώσεις, ε, εγώ θα συνεχίσω και επιπτώσεις ήδη είχα. Τώρα, το θέμα του προπολογισμού. Το έθεσαν πολλοί από εσά και πολύ σωστά. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια σειρά από εργαλεία στη διάθεσή μα. Δύο εργαλεία πιο συγκεκριμένα. Τα οποία συνδέονται με συστηματική δομική ε, δομικό μη σεβασμό των κανόνων της συνθήκης. Δύο πράγματα ε, θα γίνουν. Εάν αυτή η συστηματική παραβίαση των κανόνων των, της συνθήκης θα, υπα... θα συνεχιστεί, τότε θα υπάρξουν επιπτώσει δημοσιονομικέ. Και έχει βάλει πρόταση κομισιών για να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα συνδεθεί αυτό με το κράτο δικαίου. Και ελπίζουμε να μα υποστηρίξει το Κοινοβούλιο προ θα έχει και να πείσουμε και το Συμβούλιο να πάμε προ την κατεύθυνση αυτή. Εάν το εγκρίνουμε αυτό εν ώψη του, του επόμενου πολιτού του μεσομικού πλαισίου, σίγουρα θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Όμω, ακόμα και αν δεν το εγκρίνουμε, ε, για πόσο καιρό πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα επιτρέψουν τα χρήματά τους, τα χρήματα των φορολογουμένων να μεταφέρονται και να δίδονται σε, κράτες σε, σε κράτη-μέλη όπου χρησιμοποιούνται ε, ε, για να υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Ε, όχι και τόσο πολύ. είτε έχουμε λοιπόν αυτόν τον μηχανισμό είτε όχι, αργά ή γρήγορα, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θα πει όχι. Εμείς σταματάμε, δεν θέλουμε να το χρηματοδοτήσουμε αυτό. Καλύτερα να έχουμε τον μηχανισμό για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τους κανόνες ε, ε, στα διάφορα θεσμικά όργανα, στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν. Γι' αυτό το ζητάμε εμείς, ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε και ελπίζουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο κομμάτι είναι ευαίσθητο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο μακριά εδώ. Εάν δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο ομοιόμορφα στα κρατη αν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών, εάν δεν μπορούμε πια σε ποινικέ υποθέσει ε, να ανταλλάσσουμε ε, στοιχεία, να χρησιμοποιούμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, επειδή μπορεί να είναι βέβαιο ο δικαστή σε μία χώρα ότι ο άλλο δικαστή στην άλλη χώρα είναι ανεξάρτητο, αν καταρρεύσει και αυτό, βήμα-βήμα θα έχουμε ξανά σύνορα στην Ευρώπη. Και αναρωτιέμαι τελικά, αυτοί που μιλούν ε, για ε, ανελεύθερα καθεστώτα έχουν αντιληφθεί ότι αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσουν νέα σύνορα και αυτό θα είναι σε βάρος αυτών των χωρών, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλον. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο πληθυσμό τους. Καθόλου. Και αργά ή γρήγορα θα ξυπνήσει και ο κόσμος και θα του διορθώσει. Εγώ πραγματικά πιστεύω στην ανθεκτικότητα των Ευρωπαίων. Έχω δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει βούληση ισχυρή των πολιτών να αποτελούν μέρο μια κοινότητα αξιών όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά που θα μα οδηγήσει προ τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο μηχανισμό κράτου δικαίου την ανακοίνωση προσφορά μου προ εσά είναι να συνεχίσουμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με άλλους αυτό το διάλογο για το τι πρέπει να συμπεριληφθεί και τι όχι ε, ή τι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε προσεκτικά ε, ή διαφορετικά. Το θέμα τη ελευθερία τύπου θα είναι τεράστιο. Ε, είτε το συμπεριλάβουμε εδώ είτε κάπου αλλού. Ας γίνει μια συζήτηση Του επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια για να κάνουμε το σωστό. Επίση ε, έγινε, αναφέρθηκαν τα παραδείγματα με τα κίτρινα γυλαίκα ή στον Αμένο Βασίλειο με την παράταση τη ε, λειτουργία του Κοινοβουλίου, την αναστολή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι τελικά οι χώρε αυτέ έχουν το απαραίτητο αντίβαρο ε, που να επιτρέπουν κάποια διόρθωση. Ε, υπάρχει διαμεσολαβητή που λειτουργεί, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα βασικά. Εφόσον υπάρχουν αυτά, ό,τι και να, όποια και είναι η άποψη κάποιου για τα κίτρινα γυλαίκα ή για τα στολή λειτουργία του Κοινοβουλίου, εφόσον υπάρχει ε, ε, ε, δικαστήρι, δικαιοσύνη ανεξάρτητη, το κράτο δικαίου υπάρχει για να ανταπεξέλθει σε αυτά. Όταν δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τότε μπαίνουν ζητήματα κράτου δικαίου. Τώρα το θέμα των ΜΚΟ. Άλλο ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Έχουμε δει σε μια σειρά από χώρε, όχι μόνο αυτέ που αναφέρθηκαν, ότι περιορίζεται το πεδίο τη κοινωνία των πολιτών. Ορισμένε φορέ αυτό συμβαίνει λόγω κάποιων πολιτικών ε, βημάτων, ορισμένε φορέ γίνεται λόγω τη λιτότητα ή άλλων επιλογών που έχουν γίνει δημοσιονομικά στα κράτη-μέλη και είναι κάτι που και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Όχι για κάποιε χώρε, τι οποίε έχει κάποιο κατά νου, αλλά για όλε τι χώρε. Διότι αυτό δεν περιορίζεται σε δύο-τρία κράτη-μέλη είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα λοιπόν της κοινωνίας των πολιτών, του πεδίου που έχουν που έχει κοινωνία των πολιτών και το πώς ε, μπορεί να συμμετάσχει, είναι κάτι που μας απασχολεί. Και είναι αναπόφευκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πιο, μεγαλύτερη, περισσότερη άμεση σχέση με την κοινωνία των πολιτών στα κράτη-μέλη, εφόσον υποστηρίζουν τους στόχους ε, ε, που Έχουμε συζητήσει μια ανοιχτή κοινωνία, ποικιλόμορφη, ε, αλληλοκατανόηση. Πραγματικά πιστεύω όλο και περισσότερο ότι αυτά που ονομάζουμε παλαια παλαιά κράτη-μέλη, η σχέση με τους πολίτες έχει γίνει μια σχέση όπου οι πολίτες είναι καταναλωτές και όχι τόσο πολίτες. Οι δημόσιες αρχές δεν είναι ένα σούπερ μάρκετ που πάει κάποιος και παίρνει ό,τι θέλει. Αν ένας, πολίτ, ένας πολίτης είναι κάποιος που και αυτός συνεισφέρει, που αποτελεί μέρος ενός μηχανισμού όπου δεν έχω μόνο δικαιώματα, έχω και υποχρεώσει. απέναντι, εμένα απέναντι στους ΔΕ και απέναντι στην κοινωνία. Εάν δεν έχουμε μια ορθώ λειτουργούσα κοινωνία των πολιτών, δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μα για να καταλάβουν το πώ λειτουργεί η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό πάει πολύ πιο μακριά από τα ζητήματα κράτου δικαίου ε, σε κάποια κράτη-μέλη. Τέθηκαν κάποια ερωτήματα για το μελλοντικό κρεματορικό μου καθήκοντα, με το κρεματορικό μου χαρτοφυλάκια, χαρτοφυλάκια αυτά τα αποφασίσει η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ε, εγώ σας είπα και σας λέω εδώ ότι δεσμεύομαι να συνεχίσω τη μάχη για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τη θεμελιώδη δικαιώματα και σας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, <coughs> όπως είπε η κυρία Φόντερ Λάινεν, αυτό το θέμα θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα είναι στην πρώτη γραμμή. Για το CVM. Το CVM ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο που αφορούσε δύο κράτη-μέλη. Γιατί? Διότι όταν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 12 χρόνια δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθοράς, το κράτος δικαίου, ε, υπήρχαν ανησυχίε και αποφασίστηκε ότι το CVM θα του βοηθούσε. Βεβαίω, καταλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια απογοήτευση ότι μετά από 12 χρόνια ε, δεν έχουμε προχωρήσει τόσο όσο θα έπρεπε. Το CVM όμω διέπεται από πολύ αντικειμενικά κριτήρια. Είναι πολύ συγκεκριμένε ε, οι προποθέσει. Ε, και εφόσον πληρώνει προποθέσει, μπορούμε και να κλείσουμε το CVM. Αυτό δεν ισχύει όμω ακόμα. Εμεί θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή και με τη βουλγαρική και με τη ρουμανική κυβέρνηση για να δούμε τι πρόοδο μπορεί να σημειωθεί. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα αφορά συγκεκριμένα κράτη-μέλη, η δική μου επιθυμία είναι κάποια στιγμή αυτό να ενσωματωθεί στη γενικότερη ε, εποπτεία του κράτου δικαίου και για του 27 και 27 κράτη-μέλη, ενδεχομένω και 28. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, δεν μπορεί κανένα κράτο μέλος να είναι υπεράνω σε ό,τι αφορά αυτή την παρακολούθηση δεν υπάρχει κανένα κράτο μέλο όπου δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση του κράτου δικαίου σε κάποιου τομεί. Και ελπίζω αυτό ο μηχανισμό να συνεισφέρει ε, για να συμβεί αυτό. Βλέπω ότι κάποιοι ε, ε, έφυγαν. Α μην απαντήσω στου ανθρώπου που έχουν ήδη φύγει. Ε, ευχαριστώ πολύ. Kindly please allow me to conclude by thanking you. Σας ευχαριστούμε και να ολοκληρώσουμε με ευχαριστίες. Να συνοψίσουμε, διότι είναι μακρά η ιστορία μας, μεγάλος αριθμός ψηφισμάτων που έχει κρίνει το Ευρωκοινοβούλιο ούτως ή άλλως και υπάρχει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει έναν διεξοδικό και πλήρη μηχανισμό. Βεβαίω υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που είναι νεοεκλογέντε και νεοεκλεγήσε. Έχουν κάθε δικαίωμα να μας θυμίζουν και να μας επισημαίνουν το αρχείο των ψηφισμάτων που έχουμε γκρίνει, γιατί το γνώριζαν απ' έξω τώρα, αλλά αυτό, Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, δείχνει ότι ως πολιτικό σώμα τελικά διαθέτουμε πλειοψηφία για να στηρίξουμε και να επενέσουμε την τόλμη, την αφοσίωση, την ε, ε, ευφυΐα και την δυνατότητα να προσφέρετε και να φέρετε απτά αποτελέσματα. Παρόλο που η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδεύει προς το τέρμα της, σας ευχόμαστε κάθε τύχη το χαρτοφυλάκι που θα αναλάβετε μελλοντικά ως Επίτροπος. Καλή σας τύχη. As Vice President Timmermans waved goodbye, it will be just a minute before we resume our work with the following point of the other day, which is the presentation. Ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκινήσει η συνεδρίαση για την ΕΑΣΟ με την κυρία Γκρεκόρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ζητώ συγγνώμη από την Διευθύντρια του Γραφείου Υποστήριξης του Ασύλου, από την κυρία Γκρεκόρη. Να καθίσουμε και να συγκεντρωθούμε παρακαλώ. Μη φλιαρείτε εκεί πέρα. We thank you for that. Because we are to resume our work να συγκεντρωθούμε σιγά σιγά στη δουλειά μας παρακαλώ. Μην ψάχνουμε δικαιολογίε. Λοιπόν, θέλω να δώσω το λόγο στην ομιλήτρια για το επόμενο σημείο, την κυρία Νέα που είναι η εκτελεστική διευθύντρια της ΕΑΣΟ. Συγγνώμη σας, ε, κάναμε να περιμένετε. Είδατε όμως ότι είχαμε λόγο, είχαμε μια αρκετά θερμή συζήτηση για το κράτος δικαίου, πολύ ζωντανή συζήτηση, αυτό να λέγεται, και ίσως και διχαστική. Τέλος πάντων, συγκρουσιακή ενίοτε με τους βουλευτές. Ας περάσουμε όμως τώρα απευθείας στην παρουσίαση του έργου της ΕΑΣΟ η κυρία Γκριγκόρη ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα, φέτος μόλις, και έχει σημαντικά καθήκοντα να φέρει σε πέρας, τα οποία σχετίζονται με ένα από τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, ε, δηλαδή το σύστημα παροχής ασύλου, που είναι υπό δημιουργία. Και στο πλαίσιο της ΑΣΟ, που και αυτή ε, σιγά σιγά ε, συγκροτείται και εξελίσσεται. από το 10 και μετά να προσαρμοστεί στις νέες συντεταγμένες, ε, στο, στη νέα κατάσταση. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, έχουμε μάλιστα ορίσει τον ε, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ως εισηγητή, τον Κλοντ Μωράες. Θα ακούσουμε όμως την παρουσία σε την κυρία Νίνα Γρηγόρη και θα ακούσουμε και τι ανάγκες έχει σε δημοσιονομικά ε, από δημοσιονομικά μέτρα ή ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόβλημα ήταν η απαλλαγή. Η απαλλαγή της ΕΑΣΟ για το 2017. Το έχουμε ήδη λοιπόν συζητήσει ε, εν ώψη της ε, διαδικασίας αυτής και έχουμε τώρα εκ νέου τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω την ε, κατάσταση σε αυτή την συνεδρίαση και ήταν θερμή η συζήτηση, είπατε, ε, στο προηγούμενο σημείο της ημερησίας διάταξη. Ελπίζω ε, αντίθετα να μην βαρεθείτε σε αυτό το σημείο. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Το ΕΑΣΟ είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ένας πολύ σημαντικός εκτελεστικός οργανισμός και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα πώς ε, προχωρούμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, διότι έχουμε έναν ε, συνεχή διάλογο ως ε, υπηρεσία με όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Και είμαι προσιλωμένη σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχετε τα σχετικά στοιχεία, πληροφορίες, τις αναλύσεις που εμείς παράγουμε, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει και εσάς στη δική σας δουλειά. Όποτε λοιπόν μας χρειάζεστε, σα παρακαλώ να έρχεστε απευθείας σε επαφή μαζί μα. Στην παρουσίασή μου τώρα, καταρχάς, όπως είναι φυσικό, θα ξεκινήσω με τους ε, τρεις βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας. Ποιο είναι ο ρόλος. Βασικός ρόλος φυσικά είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στον τομέα της μετανάστευση, κυρίως όμω στον τομέα του ασύλου. Τρει βασικοί τομεί, τρία βασικά καθήκοντα, παροχή βοήθεια, ή υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή ε, του κοινού συστήματος παροχής ασύλου και πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων στον τομέα αυτό. Δεύτερον, είμαι ένα κέντρο ε, εμπειρογνωμοσύνη για ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε θέματα ασύλου. Και τρίτον, παρέχουμε πολύ συγκεκριμένη υποστήριξη στα κράτη-μέλη που είναι στο πρώτο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν ε, τις ε, αιτήσει ε, ασύλου. Να σας πω τώρα λίγο περισσότερα για το πώς έχει κατάσταση μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω θα το βρείτε ενδιαφέρον. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία εμείς περιλαμβάνουμε στις εξαμηνίες και ετήσιες εκθέσεις και αναλύσεις μας και στις ανοιχτές πηγές επίσης μπορείτε να τα βρείτε. Όταν λοιπόν συζητούμε για τη διεθνή προστασία για το άσυλο σήμερα στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι σχεδόν 338.000 αιτήσει παροχής ασύλου κατατέθηκαν το πρώτο ήμιση της φετινής χρονιάς μόλις. Και αυτό είναι το 11%, μάλλον αύξηση της ε, τάξης του 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα όμως αντίθετα μειώθηκαν. Ε, όταν ε, σήμερα μιλάμε με νούμερα βλέπουμε ότι έχουμε τέσσερις φορές λιγότερες ε, ετούντες, λιγότερους, ε, μάλλον περισσότερους λέει τώρα η κυρία Γρηγόρη. Έχουμε τέσσερις φορές δηλαδή παραπάνω ετούντες άσυλο από ό,τι έχουμε αφήξει τα εξωτερικά σύνορα. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί, πολύ περισσότεροι από που έρχονται τώρα που είναι ήδη στην και ζητούν άσυλο και τέσσερις ε, κυρίως είναι οι χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα που έχουν ε, το μεγαλύτερο όγκο αυτών των αιτήσεων. Σε ό,τι αφορά κατά κεφάλιση αιτήσεις, φυσικά έχουμε διαφορές ορισμένες από τις μικρότερες χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα ε, διακρίνονται ιδιαίτερα. Οι Σύριοι πιο πολύ, μετά οι Αφγανοί, οι Βενεζολάνοι, οι Ρακινοί και οι Νιγηριανοί οι Κολομβιανοί είναι η ε, έκτη στη σειρά. Αν τα δούμε αυτά σε μια γενικότερη παγκόσμια προοπτική για το 2018, στο EU βλέπουμε ότι πάνω από το μισό όλων των αιτήσεων ε, έχουν ε, καταγραφεί εδώ και όχι στην, στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε ε, ένα 35% περίπου ένταξη, αλλά έχουμε μεγάλες διαφορές ανάλογα με την εθνικότητα, την προέλευση. Επίσης, υποθέσει υποθέσεις όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-μέλη. 900.000 περίπου το 2018. Μισές κρεμούσε πρώτο βαθμό και οι υπόλοιπε σε δεύτερο βαθμό. Η αναλυτική προσέγγιση τόσο προσανατολίζεται στο μέλλον για την έγκαιρη προειδοποίηση και γι' αυτό χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε big data, τα μεγάλα δεδομένα και εξόριξη δεδομένων για να έχουμε ένα δίκτυ ε, και στο πλαίσιο των τριτών χωρών που αυτό μας βοήθησε, ε, βοήθησε και τα ποσοστά αναγνώρισης το 2018. Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι το EU Plus ε, μπορεί να φαίνεται ε, σταθερό, να δείχνει μια σταθερή κατάσταση ό,τι αφορά το άσυλο, πρέπει όμως να δούμε ευρύτερα ε, την κατάσταση και την εικόνα. Και τότε ξεκαθαρίζει το τοπίο και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση παρά το ότι έχουμε πολύ λιγότερου παράτυπου μετανάστε, εξακολουθούμε να έχουμε πολλέ αιτήσει παροχή ασύλου. Έχουμε σημαντικέ μετακινήσει και επανειλημμένε καταθέσει αιτήσεων. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσει και σε επιβάρυνση των αρχών των κρατών μελών. Επίση, υπάρχουν πάρα πολλέ ενστάσει και προσφυγέ ε, για την ανέρεση κάποιων αρνητικών αποφάσεων. Υπάρχουν διάφορα είδη φόρτου εργασίας ε, και φυσικά ανάλογα με την υπηκότητα ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα η τακτική και έγκαιρη ανάλυση είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και σίγουρα πρέπει να ε, το λάβουμε αυτό υπόψη για να κατανοήσουμε και την κατάσταση με το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περνάω τώρα στις βασικές μας δραστηριότητες. Όταν μιλάμε για τη στήριξη ε, που παρέχουμε στο κοινό σύστημα παροχής ασύλου. Ε, καλό είναι να ξεκινήσω με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχουμε, το οποίο αποτελείται από 24 διαφορετικές ε, συνιστώσεις, θεματικές ενότητες που χωρίζονται σε πέντε δέσμες ή ομάδες διαφορετικές και έχουμε εκπαιδεύσει ήδη 30.000 και πάνω ειδικού στον τομέα του ασύλου από όλη την Ευρώπη. Τα βασικά αυτά ε, μαθήματα, οι βασικέ θεματικέ ενότητε είναι σχεδιασμένε ώστε οι αξιωματούχοι ε, τη Ένωση να έχουν συγκεκριμένε δεξιότητε γνώση ε, στον τομέα τη διαδικασία παροχή ασύλου. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι παρακολουθούν ε, τα μαθήματά μας εν συνεχεία μπορούν να ασχοληθούν ως case officers, έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας, ε, για να διεξάγουν συνεντεύξεις με τους ετούντες και για να αξιολογούν εν συνεχεία τα στοιχεία για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Δεύτερη θεματική ενότητα. Πιο πολύ εστιάζει σε άτομα με ειδικέ ανάγκες και τεχνικές συνέντευξης που σημαίνει ότι προσπαθούμε βέβαια να εκπαιδεύσουμε τις ειδικού ε, όταν θα χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με παιδιά, με ε, αντικείμενα διακίνησης, με άτομα με ειδικές ανάγκες για θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, γενετήσια ταυτότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό και επεξεργαζόμαστε τα σχετικά τώρα για την υποδοχή αυτών των ατόμων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ειδική γνώση και σε θέματα όπως είναι το COI, η πληροφορία για την χώρα προέλευσης, ε, αποκλεισμό, υποδοχή, κανονισμός Δουβλίνου και τέλος έχουμε επιχειρησιακή κατάρτιση ε, που είναι σε συνεχή εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι οι εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη, οι οποίοι ε, θα πάνε στα κράτη πρώτης γραμμής, έχουν και μια ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να φέρουν σε πέρα στη δουλειά τους επιτόπου. Ε, πρώτο εξάμεινο του 19. Μέχρι τότε είχαν πάνω από 5.300 συμμετέχοντες στην επιχειρησιακή αυτή κατάρτιση. Τώρα, όταν μιλάμε για υποστήριξη και πρακτική συνεργασία σε θέματα ασύλου. Εδώ έχω να σας πω τα εξής. Ως φορέας που έχει εμπειρία στον τομέα αυτό, έχουμε τρία κλάστερ αν θέλετε, τρεις δέσμες ενίσχυσης πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των εμπειρογνωμόνων. Αυτό πώς γίνεται με τα λεγόμενα θεματικά δίκτυα. Δηλαδή, οι εμπειρογνώμονε, οι ειδικοί, είναι μέλο των δικτύων αυτών και συζητούν τι βέλτιστε πρακτικέ, ε, παρέχουν κατευθύνσει, καθοδήγηση και παράγουν κάποια εργαλεία για να υπάρχει κάποια αναρμόνιση των διαδικασιών ασύλου μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί ο στόχο μα τελικά είναι να φτάσουμε σε ένα κοινό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 12 τέτοια δίκτυα πρακτική ε, συνεργασία. Περιλαμβάνει και τη χαρτογράφηση των ε, καλών πρακτικών, ε, στοιχεία μετρικά και ανάπτυξη βέβαια πρακτικών οδηγιών για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην καθημερινή τους δουλειά. Πληροφορίες χώρες προέλευσης και καθοδήγηση χώρων. Αυτά είναι τα βασικά στην τρίτη δέσμη. Και ίσως ε, ο σημαντικότερος πυλώνας μας είναι οι επιχειρήσεις μας φυσικά. Τέσσερις, ε, τέσσερα επιχειρησιακά σχέδια έχουμε αυτή τη στιγμή με τα τέσσερα κράτη πρώτης γραμμής ε, που βλέπετε. Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Κύπρο. Πολύ συγκεκριμένα στην Ελλάδα παρέχουμε συγκεκριμένη υποστήριξη για να μειωθούν οι καθυστερήσεις σε πρώτο βαθμό και για τις διαδικασίες στα σύνορα με, παρου, με πληροφορίες, ε, ε, την ε, συνέντευξη και την καταχώρηση των γνώμων και από των γνωμών απόψεων και βοηθάμε και στη δεύτερη γραμμή υποδοχής, όπως τα hot spot για παράδειγμα. Στη μονάδα του Δουβλίνου της Ελλάδας παρέχουμε βοήθεια για να καθυστερήσουμε σε δεύτερο βαθμό επίσης, μάλλον για να μειωθούν σε δεύτερο βαθμό οι καθυστερήσεις. Στην Ιταλία παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, παρέχουμε πληροφορίες και έχουμε αποσπάσει ειδικό προσωπικό και παρέχουμε και άμεση επιχειρησιακή υποστήριξη στην Ιταλία, στο Κουεστούρε για παράδειγμα και στην Δαφική Επιτροπή για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές και μειώσαμε αυτές τις καθυστερήσεις κατά 50% και περισσότερο. Πολύ επικοδομητική συνεργασία μας στην Ιταλία. Στηρίζουμε επίσης τη μονάδα Δουδουβλίνου ε, και τη μονάδα για τις ε, πληροφορίες χώρες προέλευσης ε, στη Μάλτα πρώτος βαθμός ε, για την καταγραφή των απόψεων, ε, για την υποδοχή και τα λοιπά κάνουμε ό,τι μπορούμε και στην Κύπρο πρόσφατα άνοιξε το γραφείο για να έχουμε μείωση καστέρου σε πρώτο βαθμό για την υποδοχή, ε, την ευαλωτότητα και θέλουμε να δημιουργήσουμε κέντρα υποδοχή σε ασφαλείς ζώνες, κάτι που είναι αναγκαίο στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Επίσης, Πρέπει να πω φυσικά ότι πρόσφατα το γραφείο μας συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επιχειρήσεις ε, με τις λεγόμενες αποβιβάσεις ε, και τη μετεγκατάσταση ορισμένων από, αυτού ε, από αυτούς τους ανθρώπους σε άλλες χώρες. Στηρίξαμε Ιταλία, στηρίξαμε Μάλτα με πολύ συγκεκριμένη δουλειά επιτόπου όταν είχαμε αποβιβάσεις ανθρώπων στις δύο αυτές χώρες μαζί με την Κομισιόν που συντονίζει βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τα όλα εγχείρημα, έχουμε αναπτύξει το μοντέλο της Μεσίνας, όπως το λέμε. Είναι ένα μοντέλο το οποίο πιστεύουν θα βοηθήσει να εστιάσουμε κυρίως στην καταχώρηση όσων αποβιβάζονται σε Μάλτα και Ιταλία, να κάνουμε συνεταίξουν αυτά τα άτομα και έπειτα βέβαια να βοηθήσουμε και τις αρχές να εντάξουν τα άτομα αυτά στο σύστημα του Δουβλίνου. Εδώ, στο πλαίσιο του άρθρου 17 του κανονισμού του Δουβλίνου. Με αυτό το μοντέλο βοηθούμε να γίνει η λεγόμενη αντιστήχηση, matching. Και αυτοί που φτάνουν Ιταλία και Μάλτα, αρχικά, εγκαθίστανται σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Τώρα, αν να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα. 11 τέτοιες επιχειρήσεις είχαμε και βέβαια με το Ocean Viking που ήταν το τελευταίο 355 άτομα. Ο μεγαλύτερος αριθμός για φέτος μάλιστα. Όταν μιλάμε τώρα, για να σας δώσω κάποια νούμερα, για προσωπικό, ξέρετε ότι είχαμε ε, την έδρα μας στη Μάλτα. Τώρα έχουμε 292 υπαλλήλους ε, στη Βαλέτα που είναι η έδρα, τα κεντρικά. Για φέτος προβλέπουμε ότι θα έχουμε λίγο παραπάνω από 100. 390 δηλαδή ελπίζουμε να είναι στα κεντρικά μας στη Μάλτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το επόμενο έτος το προσωπικό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τη Δημοσιονομική Αρχή προβλέπονται 500 άτομα μέχρι το τέλος του 2020. Πάντα για τη Μάλτα, για τα κεντρικά, στη Βαλέτα. Ο προπολογισμό φυσικά όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως και χαίρομαι γιατί ο διάλογος ήταν πολύ επιτυχής, πολύ επικοδομητικός Άρα για το επόμενο έτος θα αυξηθεί ο προπολογισμό σε γύρω στα 139 εκατομμύρια ευρώ θα είναι μέχρι τα τέλη του 2019 και στο τέλη του 2021 ελπίζουμε να έχουμε γύρω στα 142 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό μας. Τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, είναι και τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε και με αυτό θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε την παρέμβασή μου. Και θα σας δώσω βέβαια και το μελλοντικό μας όραμα. Όλοι γνωρίζετε βέβαια ότι πρόταση για τη δημιουργία ενός οργανισμού Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Ασύλου και ο σχετικός κανονισμός είναι κομμάτι αυτής της δέσμης μέτρων ε, για το άσυλο. Εμείς δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια, η εντολή μας είναι περιορισμένη. δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αδελφό οργανισμό Frontex σε αυτά που κάνει, γιατί έχει διαφορετική εντολή. Για να είμαι πολύ συγκεκριμένη λοιπόν, όταν εμείς εργαζόμαστε και μιλά συγκεκριμένα για επιχειρήσεις επιτόπου, ενώ η Frontex μπορεί να ασχοληθεί και με την υποστήριξη ε, της μετανάστευσης ή της διαχείρισης της μετανάστευσης, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς ε, έχουμε την εντολή για το άσυλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέραν το να συντονίζουμε το έργο μας με τις άλλες υπηρεσίες. Θεσμικά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες υποστήριξης για τη διαχείριση μετανάστευσης, όπως ε, με τη Frontex με την Europol. Επίσης, Υπάρχει το λεγόμενο reserve pool, δηλαδή μια εφεδρική δεξαμενή εμπειρογνωμόνων. Δεν το έχουμε ακριβώς αυτό. Εξαρτώμεθα από άλλους, αν θα μας στείλουν τους εμπειρογνώμονες που έπειτα αναπτύσσουμε και εργάζονται για την ΕΑΣΟ στις χώρες μέλη πρώτης γραμμής. Δεν μπορώ να έχω λοιπόν παραπάνω προσωπικό από αυτό που προβλέπετε. «14% μόλις του προσωπικού είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται ε, για να μας ε, βοηθήσουν. Και δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό είναι επαρκές. Θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις βέβαια και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ενίσχυση. Κάτι άλλο πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ξεκίνησα ως εκτελεστική διευθύντρια πριν τρεις μήνες θεώρησα ότι ίσως είναι και από τις μέγιστες προτεραιότητες με τις χώρες τις οποίες ε, διεξάγουμε επιχειρήσεις δεν έχουμε ε, ολοκληρώσει τις διαδικασίες ε, φιλοξενίας hosting arrangements με την Ελλάδα ή με την Ιταλία για παράδειγμα. Δεν τα έχουμε ολοκληρώσει και αυτό είναι σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε πολύ καλή ε, συνεργασία και καλά αποτελέσματα. Δεν θέλω όμως να κλείσω με αρνητική νότα. Νομίζω ότι έχουμε ένα σαφές όραμα ως ΕΑΣΟ. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και φυσικά θέλουμε να έχουμε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Αυτό λοιπόν που επιθυμώ και εύχομαι για την ΕΑΣΟ στο μέλλον είναι τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να παραμείνει και να ε, βελτιωθεί ως ένας πρωταγωνιστής στο πλαίσιο της απαμείνησης του κοινού συστήματος ασύλου. Θα ήθελα να γίνει και να παραμείνει κέντρο ε, εμπειρογνωμοσύνης ε, σκαπανέας πρωτοπόρος για την ανταλλαγή πληροφοριών και διεξαγωγή αναλύσεων στον τομέα της μετανάστευσης και φυσικά του ασύλου. Γιατί με πραγματικέ πληροφορίες, με την πραγματική πληροφόρηση που θα πάρετε από εμά, φυσικά μπορείτε κι εσείς μετά να δημιουργήσετε πολιτική με ουσία, πολιτική με νόημα. Δεν θέλουμε με βάση ψευδείς ειδήσει να χαράσετε η πολιτική. Και γι' αυτό ελπίζω να στηριχθεί και η περαιτέρω αύξηση του προπολογισμού για αυτόν τον τομέα. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστής, μοχλός για επιχειρήσεις επιτόπου και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τις χώρες που πραγματικά μας χρειάζονται, τις χώρες προς γραμμής. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, τόσο δυναμική και με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και ενέργεια να μας προσιάζετε τον ΕΑΖΟ. Είναι καθοριστική σημασία για τη δουλειά μας ως συνομοθέτου στο, στο σώμα αυτό και για τη δουλειά της δικής μας Επιτροπής. Θα έχετε τη στήριξή μας και με όλη μας την αφοσίωση θα βοηθήσουμε να γίνει η δουλειά και να πάνε τα πράγματα μπροστά. Τώρα για την ορθότητα της διαδικασίας. Πρώτον, θα ακούσουμε την εισηγήτρια. Τον εισηγητή μάλλον, τον κύριο Κλοντ Μωράης, εισηγητή για τον κανονισμό ΕΑΣΟ. Και μετά, τους σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες. Κλοντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ κατά πολύ με όσα είπες, Χουάν. Η νέα ομάδα διοίκηση και η κυρία Γκρεγόρη έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Δεν πρόκειται για κάποια διάθεση καλοπισμού του πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Είναι ένα ντοσχέ σημαντικό και το γνωρίζω ως υπεύθυνο εισηγητής για το θέμα. Υπάρχουν ε, συνεισφορές από εμπειρότατα μέλη με την υποστήριξη και της εμπειρότατης γραμματείας και όλων των συναδέλφων. Οπότε καλό θα ήταν να συνεχίσουμε αυτού του είδους τη συνεργασία με, την, ε, με τον ΕΑΖΟ. Είστε ένας οργανισμός που λειτουργεί πλήρως πλέον και από την ε, σκοπιά της ΛΥΜΠΕ πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε με ακρίβεια και να μπορούμε να πούμε την αλήθεια ε, για το πώς ε, λειτουργεί στην πράξη ένας τέτοιος οργανισμός. Έχετε 292 υπαλλήλους σε χώρο, στον τομέα της αστυνόμευσης συγκεκριμένα, έναν από τους πιο ευαίσθητους και υπάρχει μια ποικιλία καθηκόντων που πρέπει να φέρετε εις πέρας από την διαχείριση πληροφοριών και την τήρησή τους, από αυτά που συζητάμε τώρα, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον backlog, τα γραφεία υποστήριξης αντιμετωπίζουν εδώ δυσκολίες, διότι αυτά είναι τα νέα προβλήματα με το άσυλο. Τα νέα προβλήματα που αναδύονται. Έχει λήξει, έχει εκπνεύσει μια προθεσμία και αρχίζουν να επιβάλλονται τιμωρητικές ε, τιμωρητικά μέτρα από κάποια κρατημέλη. Αυτό είναι θέμα απιστοφυλακή. Στην εμπροστοφυλακή όμως φάνηκε ξεκάθαρα και από την ε, παρουσίασή σας <clears throat> πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Είναι σαφή λοιπόν όλα αυτά. Τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Πρώτα απ' όλα το πολιτικό αδιέξοδο. και το καθήκον που έχει οποιοδήποτε εισηγητή να κάνει καλά τη δουλειά του. Θα προσπαθήσω να προωθήσω τι θέσει του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να είμαστε και σαφεί για τα νέα μέλη που βλέπουν τον τοσχέ αυτό πρώτη φορά. Ε, να είμαστε σαφεί. Είναι προτεραιότητα και για τη δική μα την ομάδα και για άλλε ομάδε. Η πολιτική όμω κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερή, ε, εφόσον δεν έχουμε πακέτο για το άσυλο. Η κατάσταση είναι επίση δύσκολη για τον επιπλέον λόγο ότι δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα έρθει να ταιριάξει το γραφείο για το άσυλο στο όλο πακέτο. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για μια γενική προσέγγιση. Η πρόταση της Επιτροπής απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, και υπάρχει και κάτι επιπλέον, ένας ακόμη ενδιασμό. Ακούμε, και θέλω να το θίξω, διότι πρέπει να ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε, ακούμε ότι η Επιτροπή μιλάει για αναστολή του Δουβλίνου και του κανονισμού του Δουβλίνου και ενδεχομένω για την όλη διαδικασία ασύλου και ενδεχομένω και για τον ίδιο τον ΕΑΣΟ. Βεβαίω θα αναλάβει σύντομα μια νέα επιτροπή τα καθήκοντά τη, αλλά καλό θα ήταν ήδη να γνωρίζουμε χοντρικά που πηγαίνουμε με όλα αυτά. Η δική μας στάση ήταν να υποστηρίξουμε τη λύση πακέτου Και πιστεύουμε ότι ο οργανισμός ΕΑΣΟ, το γραφείο για το άσυλο δηλαδή, θα πρέπει να συντεριάξει, να συνομωστεί σε αυτό το πακέτο αρμονικά. Θέλουμε να προχωρήσει πολιτικά το πακέτο αυτό για να φανεί και τι η αξία μπορεί να προσφέρει ο οργανισμό σα. Όμω το θέμα είναι θα γίνει και τι επόμενε εβδομάδε και πώ θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Τι ακριβώ θα προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον του γραφείου. Ε, δεύτερον, Έγινε χθε συζήτηση για την απαλλαγή και για την εσωτερική διαδικτύωση και οργάνωση του γραφείου. Ένα-δυο σχόλια και εδώ να πω ότι από τη σκοπιά της ΛΥΜΠΕ θα το συζητήσουμε εκτενώς βέβαια μεταξύ των μελών εδώ, αλλά πρέπει να πω ότι έγιναν πολλά θετικά βήματα όπως είπε και ο Πρόεδρος. Συναντηθήκατε επανειλημμένως με μονομένα μέλη της Επιτροπής Βεβαίω το θέμα είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, αλλά έγιναν βήματα εσωτερικώ και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε. Το αναφέρουμε διότι είναι μέρο τη διεθνωτική μα προσέγγιση και πρέπει να πω ότι θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της. Φτάνω λοιπόν και στην τρίτη μου παρατήρηση επί της ουσίας των όσων μόλις συζητήσατε δηλαδή οι τωρινέ δυσκολίε του οργανισμού. Πιστεύω ότι είναι τεράστιε. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξής. Και με αυτό να ολοκληρώσω. Το γραφείο του ασύλου πρέπει να λειτουργεί ευθύς, να λειτουργήσει ευθύς αμέσως με τον αριθμό των 292 υπαλλήλων και άσχετα με την πολιτική κατάσταση που στην οποία βρισκόμαστε και με την εκκρεμότητα του πακέτου ασύλου που ακόμη δεν έχουμε. Κατά την άποψή μου πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό που κάνετε τώρα για να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην ε, νέα, την ανανεωμένη προστεθέμενη αξία που μπορεί να έχετε. Πρέπει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δυστυχώς προβλέψει έναν ε, πολύ περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, μη ρεαλιστικό, για να ασχοληθεί με ένα τόσο τεράστιο όγκο δουλειά. Πρέπει όμως τα γραφεία για το άσυλο να λειτουργήσουν ε, γρήγορα και αποτελεσματικά και νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής θέλουν να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Ξεκινάμε αμέσως. Σήμερα, τώρα Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε και το πολιτικό αδιέξοδο. Θα πάψω εδώ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο διατόν συντομότερα. Δεν βλέπω να είναι εδώ και ο εισηγητής από το ΕΛΚ. Ο κύριος Τομαστόμπι δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Να περάσουμε στο σκιώδη εισηγητής από τους Renew. Η κυρία Σάρα Ντόναθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο εάν γίνεται διότι είμαστε κάπως πίσω στο χρόνο δυστυχώς is the minute which the next ε, hearing should be getting. Κανονικά θα πρέπει να αρχίσει τώρα η επόμενη ακρόαση με την διευθυντή της Ιγιολίσσα. Βεβαίω, προφανώ ε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την μέσα διάταξη. Ε, βοηθήστε μα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά σύντομη. Ευχαριστώ. Με ευχαριστήσω την κυρία Γκρέγκορη για την, ε, για την ε, σύνοψη των εργασιών σας. Σας ευχαριστώ και για το έργο σας ε, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να απαντούν στις μεγάλες, στη μεγάλη πνευματική πίεση που υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι φεύγουν από εμπόλεμε ζώνε και κινδυνεύουν για τη ζωή του και δεν γίνεται σεβαστή ούτε το δικαίωμα στη ζωή του, ενώ το Συμβούλιο δεν μπορεί ε, να βρει άκρη. Πώ αξιολογείτε τα κράτη-μέλη ε, και τι δυνατότητέ του να αντιμετωπίσουν τι μεταναστευτικέ ροέ, Έχετε σημειώσει κάποια βελτίωση από αυτού το τελευταίο έτο ε, και πού είναι τα μεγαλύτερα κενά κατά τη γνώμη σα. Και το άλλο ερώτημά μου είναι το εξή. Σε μια κατάσταση κρίσης άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες, ε, παιδιά, ε, μειοψηφίες είναι πιο ευάλωτα απέναντι στις διακρίσεις, απέναντι στη βία, απέναντι στην δίωξη. Ε, ε πώς εσείς αξιολογείτε τις ειδικέ ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Ναι, να είστε σύντομοι για να μας βοηθήσετε. Και τώρα για τους πράσινους και ως συγητής ο κύριος Ντάμιαν Μποσλάγκερ είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους αδέλφους να σας συγχαρώ για το έργο σας για τα ζητήματα αυτά ε, και χθες ε, στην Επιτροπή ε, Κοντ είδαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Θα ήθελα και εγώ όπως και οι συνάδελφοι να πω ότι βεβαίως είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα με το πακέτο αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα πριν ε, δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έχετε μιλήσει για ενίσχυση της υπηρεσίας σας, είναι αυτό απαραίτητο ε, για να μπορέσετε να διαβρύνετε τις δραστηριότητές σας. Οι υπηρεσίε αυτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα τη και του ασύλου είναι εξαιρετικά σημαντικέ, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή και αυτό το ζητάμε εδώ και καιρό. Ένα ερώτημα από την ομάδα μου για τη διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις από, για τις χώρες προέλευσης. Ε, μπορείτε να μας πείτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις ε, και επίσης λίγο πιο προσωπικά ε, εσείς ε, πέρα από αυτά τα οποία αναφέρθηκα για το πακέτο τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή για να σας υποστηρίξει. Από τους ID παρακαλώ, την ECR, υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο, δεν είναι εδώ, και από την ΚΟΕ. Ο Μικελάχελ Ουρμπάν δεν είναι εδώ επίσης. Ωραία, αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση τη συζήτηση και με τους υπόλοιπου ομιλητές. Παρακαλώ κυρία πρόεδρο η Μαΐτε. Ευχαριστώ πολύ πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Είναι προφανές ότι λείπει το πακέτο για το άσυλο, λείπει η νομική βάση, λείπουν πόροι. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς μπορείτε να κάνετε αναλύσει, αλλά στις αναλύσεις σας να ζητάτε και κάποια πράγματα. Έχετε πάει στη Λέσβο, έχετε πάει στη Μόρια. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι εκεί ε, ουσιαστικά κατασκευάζουμε ε, ψυχικά τραύματα στους ανθρώπους. Ε, οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές. Είναι μια πραγματική κόλαση για τους ανθρώπους εκεί και δεν πληρείς προϋποθέσεις ε, ενός hot spot. Θα ήθελα λοιπόν στην ανάλυση σας να πείτε ότι σε περιοχές όπως η Μόρια, η Μόρια πρέπει να κλείσει. Πήγα το 2016, πήγα και φέτος και είναι πραγματικά κάτι αβάσταχτο. Μπόρεσα ε, να, θα, θα να μπορέσω να συναντήσω κάποιον από, από την ε, αντιπροσωπεία σας επίσης. Ο Παδάκης έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο hot spot στην Ελλάδα, αναφέρθηκε και η Μόρια, είναι απαράδεκτη μέσα από την αντιδραστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την οδηγία για το γεωγραφικό περιορισμό που είναι εκρηκτική η κατάσταση και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία σε συνέχεια αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει την κλιμάκωση του αυταρχισμού με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση των δευτεροβάθμιων επιτροπών και του δικαιώματο προσφυγή στου ετούντε άσυλο. Παράλληλα, συζητιέται και να αφαιρεθεί από τι ευάλωτε ομάδε ετούντων άσυλο η περίπτωση των προσώπων με σύνδρομο μετατραυματικού στρε, με το αιτιολογικό το απαράδεκτο ότι ε, το επικαλούνται συχνά οι ετούντε. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για περιφρόρηση των ειδικών αναγκών των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μετά από δυσκολία, μετά από επώδυνα σκληρά ταξίδια παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή των ίδιων και των παιδιών τους. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν πώς τοποθετήστε σε αυτά τα ζητήματα και στο γεγονός ότι το πρόβλημα δεν είναι η σύντμηση των προθεσμιών και των σταδίων της λεγόμενης ταχύρυθμης διαδικασίας εξέτασης ασύλου, αλλά η ουσία είναι να προσληφθεί παραπάνω προσωπικό, εμείς λέμε και από κρατικού υπαλλήλους που να κάνουν αυτή τη δουλειά και σωστά και γρήγορα. Euh, Κυρία Κλέρ, ευχαριστούμε. Κυρία Εκτελεστική Διευθύντρια, ευχαριστούμε πολύ για την ε, σκληρή σας δουλειά και την δράση σας. Χρειαζόμαστε μέτρα για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, ιδίω ω προ τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου και των ε, ροών. Μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Έχετε στοιχεία για την εσωτερική κυκλοφορία, το πώς μετακινούνται οι αιτούντες άσυλο στην περιοχή μου, βλέπουμε ότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχει πολλοί κόσμος που φτάνει στην Ιταλία, αλλά υποβάλλει αίτηση στη Γαλλία. Κυρία Στρίκ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Καταλαβαίνω την απογοήτευση του Άσο. Πρέπει να περιμένετε νομοθετικό πακέτο, ενώ οι αιτήσει συσσωρεύονται. Εγείρονται όμως και κάποια άλλα ερωτήματα για τα όρια των τωρινών αρμοδιοτήτων του ΕΑΣΟ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σωστή εκτίμηση α, για το τι γίνεται με τα hot spot και το τι αποφάσεις λαμβάνονται. Δηλαδή, στην Ελλάδα, ας πούμε, η ΕΑΣΟ κάνει κάποιες συστάσεις. Τι αποφάσεις παίρνουν τελικά όμως οι Έλληνες υπάλληλοι και αξιωματούχοι. Οι συμβουλές μεταφράζονται σε πράξη, εκτελούνται από τους ε, εθνικούς υπαλλήλους, διότι υποθέτω ότι στο τέλος θα μας απασχολήσει και η διάσταση της λογοδοσίας. Ποιος είναι υπεύθυνο. Μπορείτε λίγο να το εξηγήσετε πώς το ε, εντοπίζετε το θέμα και πώς τη λύση προβλέπετε. Λοιπόν, ε, και πάλι έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον διευθυντή της Ιουλίζα. Ε, περιμένει η διευθύντρια της Ιουλίζα περιμένει το ραντεβού. Θα πρέπει να βιαστούμε, αλλά παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε, κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακολούθησα τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του κανονισμού ΕΑΖΟ και αναθεώρησης του κανονισμού ΕΑΖΟ στην περασμένη θητεία ως ε, σχεδόν εισηγήτρια. Ασχολήθηκα και με αυτό και με τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν, συναποτελούν το πακέτο για το άσυλο. Πιστεύω ότι το σύστημα της Ευρώπης για το άσυλο θα πρέπει να έχει ένα πλήρες φάσμα μέτρων. Έχουμε καθυστερήσει όμως. Ελπίζουμε με την ανάληψη καθηκόντων από την Νέα Επιτροπή να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μεταρρυθμιστεί το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Μα βοηθήσατε πολύ στην Ιταλία για να μειώσουμε το χρόνο εξέταση τη κάθε και είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος προσφέρει υποστηρικτική δουλειά, την υποστήριξή της στις ε, χώρες και τους φορείς τους, ιδίως όταν βρισκόνται στα σύνορα, για να μπορούν να αποδεχτούν σωστά τους ετούντες άσυλο. Ω προ το κείμενο για την ΑΖΟ που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ προσωπικά είχα κάποιε επικριτικέ παρατηρήσει, ιδίω για την κύρωση που προβλεπόταν. Να σταματήσουν να λειτουργούν κάποια εσωτερικά ε, σύνορα, εφόσον δεν γίνονται σεβαστές κάποιες διαδικασίες που προβλέπουν οι συστάσεις της ΕΑΣΟ. Αυτό όμως για τις δευτερογενείς μετακινήσεις είναι προβληματικό, το είπε και η συνάδελφος Κελέρ. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα πραγματικό, ένα αληθινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, να υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο για το άσυλο θα ήταν πολύ ωραίο, είναι σίγουρα πρόημο να το συζητάμε τώρα και είναι απλώ μια υπόθεση για το μέλλον, αλλά ωραίο θα ήταν να υπήρχε αμοιβαία αναγνώριση από όλα τα κατημέλη του δικαιώματο στο άσυλο και του κράτου του δικαίου. ώστε να μην δημιουργούνται ανταγωνισμοί μεταξύ κρατών μελών, να μην υπάρχουν προβλήματα λόγω των δευτερογενών μετακινήσεων και όσοι αιτούνται άσυλο να αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτοι σε όλη την επικράτεια τη Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Σάντο. Ε, ζητήσατε το λόγο, αλλά νομίζω έχετε την ευγενή καλοσύνη να ε, παρατηθείτε το δικαίωμα σα να παρέμβετε, διότι έχουμε και τον διευθυντή, τη διευθύντρια Γιουλίζα που περιμένει. Παρακαλώ, κυρία Γκρεγόρη, να απαντήσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ολοκληρώσουμε γέρο την ημερήσια διάταξη τη σημερινή πρωινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ και ευχαριστώ για τι θετικέ σα ε, διδράσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι από τους βασικούς μας υποστηρικτές και εταίρους. Για να συνοψίζω λοιπόν, πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, αλλά θα μιλήσω πολύ γρήγορα, Πρόεδρε. Κουράγιο. Το θέμα της απαλλαγής 2007. Πρέπει να το θέσω. Κάποιοι από εσά δεν ήσασταν στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, αλλά υπάρχουν τεράστιες ε, αλληλεπιδράσει και προεκτάσει των όσων συμβαίνουν εδώ και τη δουλειά τη σε σχέση με τη δουλειά τη Κόντ. Τα είπε και ο κύριο Σαβάρμα. Σίγουρα θα σα υποβάλει την σχετική έκθεση, αλλά πρέπει να πω εδώ ότι εγώ έχω αναλάβει το νεάζο εδώ και τρει μήνε. Έχω εργαστεί στη μετανάστευση και στο άσυλο όλη μου τη, τη ζωή. Αλλά έχω αναλάβει τη διεύθυνση του ΑΖΟ εδώ και τρει μήνε. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανεί το γιατί τώρα δεν γίνονται όλα όπως πρέπει. Έγιναν και το 16 και το 17 τα ίδια. Δεν θα πάρουμε απαλλαγή, διότι της έκθεσης ε, του Όλαφ και όσων έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί τώρα ε, δημιουργεί πρόβλημα στο δικό μου τον οργανισμό, στη δική μου τη φήμη και τη δική μας τη φήμη του οργανισμού μας. Πλήττει τις βασικές μας αξίες διότι έχουμε λειτουργήσει βάσει όλων των κανόνων χρηστή δημοσιονομική διαχείρισης και όλων των εσωτερικών κανόνων. Δίνουμε μεγάλο αγώνα για να σεβαστούμε όλες τις συστάσει, τις συστάσει του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Έχουμε επιπλέον project, έχουμε αυστηρότατα μέτρα τα έχουμε δει με τους υπαλλήλου μας και με, την, ε, ε, με το Διοικητικό Συμβούλιο για, την, ε, για τις προσλήψεις, για τις δημόσιες προμήθειες, όλα. Όταν λοιπόν ψηφίσατε για την απαλλαγή, να έχετε κατά νου ότι είναι και θέμα εμπιστοσύνη. Είναι θέμα του πώς θα ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη με τον οργανισμό μας. Για τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την αποτίμηση της ικανότητας των κρατών μελών να διεκπαιρεώσουν τις αιτήσει ασύλου και τις ειδικέ ανάγκες των παιδιών ή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ναι, έχουμε πληροφορίες για τις ε, Το παρακολουθούμε σε ξαμηνιαία βάση με σχετικές εκθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να αξιολογούμε και να αποτιμούμε πλήρως. Δεν έχουμε τέτοια εντολή. Μπορούμε απλώς να προσφέρουμε πληροφορίες εσάς με την νέα εντολή, αυτό που είπε και ο εισηγητή σα, ο, παρακο... ο μηχανισμός παρακολούθησης θα επιτρέπει να διοργανωθούμε κι αλλιώ στο εσωτερικό του οργανισμού. Αν πάρουμε λοιπόν εντολή για αποτίμηση και για αξιολόγηση, εντάξει, μπορεί να γίνει. Θα μπορούμε να βάλουμε και βαθμού στις χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε που πάνε άσχημα τα πράγματα, ποιοι είναι οι λόγοι και τι υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε εμεί. Αλλά σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το για τις εκθέσεις για τις χώρες προέλευσης. Το είπε η συζητήτρια. Και τις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι σαφές ότι είναι βασικό αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινό σύστημα ασύλου αν τα κράτη-μέλη δεν αποφασίσουν ε, με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Και με δεδομένε τι ίδιε πληροφορίε. Οι πληροφορίε λοιπόν για τι χώρε προέλευση και οι εκθέσει που τι περιλαμβάνουν πρέπει να συντάσσονται σε συνεργασία με εμπειρογνώμονε των κρατών μελών και τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΙΕ για του πρόσφυγε. Είναι τεράστιο δίκτυο αυτό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να συγκεντρωθούν ε, μαζί για να καταλήξουν, να επεξεργαστούν και να συμπιλήσουν τα σχετικά στοιχεία. Οι εκθέσει λοιπόν αυτέ είναι πολύτιμε για όλου του υπεύθυνου λήψη αποφάσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδάλω δεν θα έχουμε κοινό σύστημα ασύλου. Και εδώ να πάω πάλι στην ερώτηση για την κατάσταση στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ιδίω στην Ελλάδα. Εντάξει, η ΕΑΖΟ κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει με τις διαδικασίες, αλλά οι υποδομές ε, υποδοχής είναι στα χέρια των κρατών Εδώ προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς ζώνες εντός των χώρων υποδοχής και προσπαθούμε να προβλέψουμε ειδικέ διαδικασίες για τα παιδιά για τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες εντός των χώρων της υποδοχή, αλλά δεν είναι στα χέρια μας οι χώροι αυτοί. Εκεί αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε από τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα με την Ελλάδα. Όμως ο στόχος μας είναι να έχουμε ταχείες ε, και εύληπτε διαδικασίε. Πάω και στι δευτερογενεί μετακινήσει τώρα. Σε συνεργασία με την Frontex και την Europol, ο ΕΑΖΟ ε, έχει ολοκληρώσει μια πολύ καλή ανάλυση για το τι γίνεται με τι δευτερογενεί μετακινήσει. Υπάρχουν εκεί κάποια νέα στοιχεία. Φυσικά αυτό επηρεάζει την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε όλα τα κατημέλια. Πρέπει κάποιος να περιμένει για απόφαση για τεράστιο χρονικό διάστημα σε κάποιο κράτο μέλο. και είναι μπλοκαρισμένα εντωμεταξύ τα ατομικά δικαιώματα, προφανώς θες να μετακινηθείς κάπου αλλού. Έτσι προκαλούνται πολλές δευτερογενείς μετακινήσεις. Και εδώ θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για τις διάφορες, ε, τα διάφορα κλεισίματα σύνορων που παρατηρούμε, αλλά και για το πώς θα πάμε σε μια σύγκληση για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των κρατών μελών που δίνουν ε, δικαίωμα και ηθαγένεια μιας χώρας, ώστε να είναι παρόμοια. Ας πούμε τώρα το Αφγανιστάν, εθνικότητα του Αφγανιστάν. έτσι στην Ευρώπη, κάποια κρατημέλη έχουν κατά 60% θετική απόφαση για τέτοιες ε, αιτήσει. Σε κάποια άλλα είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Έτσι προκαλούνται πολλές δευτερογενείς μετακινήσεις. Για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή και ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε. Ελπίζω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μας επισκεφθεί ξανά. Είστε όλοι προσκεκλημένοι διαρκώς. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή τύχη. Καλή αρχή στη νέα θητεία, στην ερχόμενη πενταετία δηλαδή, με μπόλικη δουλειά και σε ό,τι αφορά το σύστημα ασύλου δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο για την Επιτροπή Λίμπε. Η κατάσταση πραγματικά είναι δραματική, είναι τραγική και μας στενοχωρεί βαθιά. Πρέπει από όλους μας να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα γίνει. Θα σταθούμε στο πλευρό σας. But you see, we got the director of EULISA ready to go. Here's the following point. Please, Director Garkov of EULISA. Παρακαλώ, κύριε Γκάρκοφ, η Γιουλίζα. Kindly excuse us for the delay. Να μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. We welcome right away Director ο κύριος Γκάρκοφ, ο τελεστικός διευθυντής ε, του EU Λίσα είναι εδώ για την επιχειρησιακή διαχείριση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας στον τομέα δικαιοσύνης, ε, δικαιοσύνης ε, και ελευθεριών και του σχετικού οργανισμού ΦΡΑ. Ο πρώτος κανονισμός εγκρίθηκε το 2011, τέθηκε σε ισχύ το 2012, ήμουν εδώ, όταν δώσαμε έτσι και ένα σπροξηματάκι γιατί θέλαμε να έχουμε έναν οργανισμό που θα χειρίζεται ε, συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας ε, στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας οσύνης. Και υπάρχουν τώρα πολλές νέες προκλήσεις. Γι' αυτό και έχουμε διευρύνει την εντολή του οργανισμού από το 2018. και έχει πλέον ένα μεγαλύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων για να αντιμετωπίζει τα θέματα της διαλειτουργικότητας που μας έχει γίνει ψύχωση τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει την ασφάλεια κάτι που φυσικά μας ενδιαφέρει γιατί μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά έχουμε και τα ζητήματα της ιδιωτικότητας, της ψευτικότητας δεδομένων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ακαιρεότητας, δικαιώματα πολίτη, προσώπου. Όλα αυτά τα κατοχυρώνει ο χάρτης ε, των δικαιωμάτων και ο οργανισμός ή Λίσα. πρέπει να εφαρμόσει και να χρησιμοποιήσει και τα εργαλεία της Γιούροντα και άλλων. Α, και το αιτία, το έκρης, σύστημα εισόδων-εξόδου. Κύριε Γκάρκοφ, καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε και ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει με υπέρβαση δυστυχώς ωραρίου σε κανένα μισάωρο. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει όταν βάζουμε όλα στις ε, υπηρεσίες εδώ στην Μερσιά Διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ να σας συγχαρώ που εκλεγήκατε πρώτα απ' όλα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που έχετε να επιτελέσετε. Η ίδρυση αυτού του οργανισμού, ιδίως ε, μετά τις νέες προτάσεις που συζητήσατε πέρυσι για νέα συστήματα, θέλουμε να έχουμε ανοιχτές ειλικρινείς σχέσεις με την Επιτροπή σας, ε, όπως είχαμε και κατά το παρελθόν για να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Θα συνεχίσουμε ακριβώς με αυτήν την υποστήριξη και στη Νέα Θητεία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε στο κέντρο της Ένωσης ε, το χώρο Σέγγεν, που θεωρείται από τους Ευρωπαίους πολίτες ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ε, ο χώρος ελευθερίας ασφάλειας δικαιοσύνης ε, ε, επιτρέπει σε πάνω από 400 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ταξιδεύουν χωρίς ε, ελέγχου στα σύνορα, αλλά να νιώθουν επίσης και προστατευμένοι, ασφαλείς. Γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα ε, και επίσης δημιουργήθηκαν σύντο χρόνο και συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας. είναι αυτά τα συστήματα, η διαλειτουργικότητά τους και η επιχειρησιακή τους ε, δυνατότητα που είναι και λόγος του ύπαρξης του Ήγιου e Λίσσα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού του αναλάβαμε καθήκοντα, δείξαμε ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συμβάλλουμε στην λειτουργία του χώρου και στηρίζουμε την εφαρμογή των πολιτικών στον τομέα πολιτικής διαχείρισης συνόρων, μετανάστευση ασύλου και έχουμε παράσχει συνεχώς αξιόπιστες υπηρεσίες μέσω των συστημάτων όπως είναι το VIS, το SIS και το Eurodac. Το 2018 η διαθεσιμότητα των συστημάτων αυτών ήταν σχεδόν 100% και 96% των κρατών μελών ήταν ικανοποιημένα, πολύ ικανοποιημένα με τον τρόπο που εφαρμόζαμε την εντολή μας. Ο ρόλος ε, του EU ε, αυξήθηκε και θα διευρύνεται όλο και περισσότερο. Και για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των κρατών μελών και τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, έχουμε πλέον από τις 11 Δεκεμβρίου του 2018 μια νέα εντολή, ενισχυμένη εντολή, που δίνει περισσότερο ρόλους και αρμοδιότητες ε, στον οργανισμό μας για τη διαχείριση δεδομένων, έρευνα, πιλωτικά προγράμματα, τεχνικά πρότυπα και ad hoc υποστήριξη στα κράτη-μέλη και άλλες βέβαια και στην Κομισιόν. Μπορεί δηλαδή πλέον να στηρίξει τα κράτη-μέλη και σε περίπτωση κρίσης μεταναστευτικής, ε, κρίσης ασφάλειας ή να τις αναθέσει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να λειτουργήσει ε, κάποιες κοινέ συνιστώσεις IT. Ε, Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, αλλά οι διερμηνείς λένε ότι πρέπει να επιβραδύνεται λίγο. Ναι, απλά προσπαθώ κι εγώ να μην υπερβώ το χρόνο. Παρέχει και τεχνική κατάρτιση στα κρατημέλη ο Ιουλίσσα. Το 2018 ήταν πάνω από 40 τα διαφορετικά αυτά μαθήματα και θα αυξηθούν με τη διεύθυνση εντολή και με την εφαρμογή των νέων αυτών συστημάτων. Επίσης, καλό είναι να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της νέας εντολής του οργανισμού μας έχουμε μια διτή πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε βασικές μας δραστηριότητες και επιχειρήσεις, το σύστημα αυτό, ΣΥΣ, ΒΙΣ και Eurodac να είναι επιχειρησιακά στα κράτη. Απ' την άλλη όμως πρέπει όλο και περισσότερο να συνεισφέρουμε για, στην υπηρεσία των κρατών μελών και των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό μας για το 2018 210 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών και 93 εκατομμύρια σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Μεγάλο ποσοστό εφαρμογή των αναλήψεων υποχρεώσεων 99,5% 100% δε εκτέλεση των πληρωμών. Επίσης στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα δείτε ότι έχουμε ποσοστό εφαρμογής ε, της τάξης 90% και 162 ήταν πλήρως μέλη του προσωπικού, 122 είναι προσωρινοί, 31 συμβασιούχοι και 9 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμες. Τέλει 18 αυτά τα στοιχεία. Ανεξαρτήτως ε, του γεγονός ότι αυξάνεται η ζήτηση, έχουμε χαμηλή ανακύκλωση, 5% στο προσωπικό μας. Τώρα, να σας πω κάποια πράγματα για τα συστήματα αυτά που τόσο ενδιαφέρουν. Το ΣΥΣ είναι το πιο σημαντικό γιατί παρέχει περιχειρησιακή υποστήριξη αρχέ επιβολή τη νομοθεσία, στου συνοριοφύλακε, στου αρμόδιου για τη μετανάστευση, το άσυλο και του ε, δικαστικού εμπειρογνώμονε. Βιομετρικές ικανότητε έχουν πλέον προσαρμοστεί, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε στο σύστημα τα βιομετρικά δεδομένα για να εντοπίζουμε τους εγκληματίες, τους διάφορους. Αυτό έχει βελτιώσει την ακρίβεια και μέχρι το 2020 θα πρέπει όλα τα κρατημέλη να να χρησιμοποιούν αυτέ τις δυνατότητες. Το 2018 επίση ξεκινήσαμε την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Το 2018 6 δις ήταν οι προσβάσεις στο σύστημα. Πάνω από 60 εκατομμύριο ήταν η, τα alert την ημέρα. Ε, 82 εκατομμύρια είναι αποθηκευμένα ε, στο σύστημα. 732 hit τη μέρα. Διπλάσια τα στοιχεία σε σχέση με το 14. Το ίδιο με το VIS, που είναι η βασική πλατφόρμα για την εφαρμογή της κοινή ε, πολιτικής για τις θεωρήσεις. Το χρησιμοποιούν οι συνοριοφύλακε στα εξωτερικά σύνορα για να ελέγχουν του υπηκό των χωρών που έχουν βίζα στα χέρια του. Θέλουμε να το βελτιώσουμε αυτό το σύστημα ώστε να είναι κατάλληλο προσαρμοσμένο για το μέλλον. Ιδίω για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτού του συστήματο και του συστήματο εισόδων-εξόδων. που απαιτεί νομική βάση. Τα νούμερα δείχνουν τα πράγματα. Πάνω από 240 εκατομμύρια επιχειρήσεις το 2018. Πάνω από 64 εκατομμύριο αιτήσει θεωρήσεις. Και πάνω από 60 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα. Και το μέσος όρος των ελέγχων στα σύνορα μέσω του συστήματος είναι 3,7 εκατομμύρια τους τελευταίους μήνες. Eurodac επίσης, βασική πλατφόρμα για την εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση για την αναδιατυπωμένη πρόταση για το Eurodac, για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εργαλειοθήκη για να βλέπουμε δευτερογενείς μετακινήσεις, να ε, διευκολύνουμε την μετεγκατάσταση και να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Διευθύντρια Τεάσο για τις τάσεις. Μετά ε, την, το ταβάνι που πιάσαμε το 2015 πλέον κατεβαίνουμε. Ε, το 2018 ήταν πάνω από, μάλλον λιγότερο από ένα εκατομμύριο οι δράσεις. Και παρότι βλέπουμε να το χρησιμοποιεί πολύ ε, το σύστημα αυτό, η Ένωση, τα κράτη-μέλη τη σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεις. Τι έγινε τώρα στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Έγινε μια πολύ εκτενή συζήτηση για να εντοπιστούν κενά στην ασφάλεια και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και είχαμε μια νέα αρχιτεκτονική, η οποία ορίστηκε για τη λειτουργικότητα των νέων και για όσα θα δημιουργηθούν. Το EU-LISA προχωρά και με το αιτίας. Έχουμε αναβαθμίσει και το ΒΙΣ και έτσι θα έχουμε σύγχρονο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, μια κοινή πλατφόρμα για την ε, έρευνα των τρίτων υπηκόων, χωρίς να ε, επιβαρύνουμε τους ε, καλόπιστους ταξιδιώτες. Επίσης θα έχουμε συγκέντρωση στοιχείων για καταδίκες υπηκών τριτών χωρών. Θα δημιουργήσουμε όμως και θα αναπτύσσουμε τη νέα αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητα. Μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτή η διαλειτουργικότητα θα είναι το θεμέλιο νέας ευέλικτης ε, μοντέρνας αρχιτεκτονικής που θα βοηθά τις αρχές των κρατών μελών για να έχουν όταν τις χρειάζονται τις πληροφορίες που θέλουν. Η λειτουργικότητα και η σχετική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει βασικά, βασικούς δομικούς, ε, δομικά στοιχεία για να μην μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδή ή πλαστή ταυτότητα οι εγκληματίε. Θα ελέγχω τι πολλαπλέ ταυτότητε. Έχουμε επίση το βιομετρικό σύστημα που θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση με τη χρήση βιομετρικών πληροφοριών, ακριβέστατων και θα ελέγχουμε τις βάσεις δεδομένων επίκαιρα, εγκαίρα συγγνώμη, και αποτελεσματικά σεβόμενοι τα δικαιώματα πρόσβασης και με σεβασμό στους κανόνες των διαφόρων νομικών μέσων. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω. Για να σας πω ότι σε ό,τι αφορά αυτά τα συστήματα εισόδες, εξόδου, διαλειτουργικότητα, ε, πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Αλλά έχουμε και άλλα σημαντικά στοιχεία για το Στρασβούργο, παραδείγματος, να έχουμε το επιχειρησιακό μας κέντρο εκεί. Τα νέα μοντέλα και μονάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν. Έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θα κάνουμε πιο ισχυρή και πιο ασφαλή την Ευρώπη. Και στην ψηφιοποίηση του τομέα της δικαιοσύνης θα διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο. Εκεί ίσως ε, θα υπάρξουν και νέα καθήκοντα που θα μας ανατεθούν για την ανταλλαγή δικαστικών πληροφοριών ή κόντεξ. Το βλέπουμε και στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου για συνήθως Εσωτερικών Υποθέσεων και όλα αυτά βέβαια. Θα πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ των καθηκόντων που μας έχουν ανατεθεί και των πόρων οικονομικών και ανθρώπινων που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ιδίως ε, κρίσιμο είναι το νέο πολιετές νοσομικό πλαίσιο δεν υπάρχουν περιθώρια λιγμών κάτω από την πρόταση της Κομισιόν για το νέο πι. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας πλήρως τα καθήκοντά μας. Επίσης, πιστεύουμε ότι στο νέο πι υπάρχουν περιθώρια λιγμών στον ε, τίτλο, στον τομέα 4. Αν γίνει καλύτερη διανομή των κονδυλίων θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέγεθος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Όλα εξαρτώνται και από τις διαπραγματεύσεις για κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις αίτιας, ε, ε, βίς ε, και πολλά άλλα. Η στελέχωση κάτι είναι, κάτι, είναι κάτι ακόμη σημαντικό για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα τις νέες ε, ευθύνες που έχουμε στο πλαίσιο της διευρυμένης εντολής. Όπως είπα, είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το έργο της δικής σας Επιτροπής, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Να παρακολουθούμε λοιπόν ε, την εφαρμογή των μέτρων που έχουμε διεγκρίνει, εν αναμονή και των νέων. Τέλος. Ο οργανισμός μας ε, είναι πρόθυμος να απαντήσει οποιοδήποτε ερώτημα, να ανταποκριθεί οποιοδήποτε έτοιμο και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση. Σε ευχαριστούμε, Κρούμ Γκάρκοφ, διευθυντή της Ήταν τεράστια η μέρα μας. Ξεκινήσαμε ρωτήσουμε το πρωί με Και η φυσική κόπωση είναι αντιστρόφως ανάλογη της πολιτικής αφοσίωσης και της προσήλωσης που έχουμε στους ίδιους σκοπούς με εσά και του οργανισμού σας, όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Να υπολογίζετε σε μας και μπορείτε να βασίζετε στην υποστήριξή μας. Προσπαθήστε τώρα να Περιορίστε το χρόνο των ερωταπαντήσεων, διότι είχαμε προβλέψει ε, διάρκεια της συνεδρίασης ίσως στις 12 και 45. Εφόσον λοιπόν ξεπεράσουμε αυτό το όριο, πρώτον θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε επιπλέον λεπτά από τους διερμηνείς μας και θα τους ευχαριστήσουμε ευγενικά αν μας τα παραχωρήσουν και μετά θα χρειαστεί να μιλήσουμε αγγλικά. Είναι ο δεύτερος πόρος που έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε να συνεννοηθούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λέναρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Διευθυντά. Είναι πολύ ευχαριστώ να σας βλέπουμε εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια είχατε πολλή δουλειά. Η ο ΕΑΖΟ έχει αναλάβει τεράστιες ευθύνες ως κεντρικός πυλώνα του αρχιτεκτονήματος ασφάλεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη δουλειά σα. Δεν έχουμε μονή με την διαλειτουργικότητα, απλώ με πολύ υγιή τρόπο το αντιμετωπίζουμε και το παρακολουθούμε στενά. Είναι αυξημένε οι απαιτήσει ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι απλώ με την συλλογή περισσότερων δεδομένων, απλώ πρέπει η χρήση των δεδομένων που κάνουμε να είναι πιο ε, αποτελεσματική κυρίως για να ε, βελτιώνουμε την προστασία του ιδιωτικού βίου των πολιτών. Ε, αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής κίνηση και ανυπομονούμε για την σωστή ε, θέση σε ισχύ και εφαρμογή του σχετικού κανονισμού. Επίσης, μερικές ερωτήσεις. Αναφέρατε κάποια νομοθετικά ντοσιέ που θα πρέπει να προωθηθούν, όπως το Eurodac και τις αλλαγές στο Ίκρες και στο ΙΤΙΑΣ τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στη διαλειτουργικότητα εάν δεν έχουμε γέρος τους επικυροποιημένους κανονισμούς γρήγορα. Πώς θα επηρεάσει τη δουλειά σας στην διαλειτουργικότητα. Αναφέρατε και το σύστημα ΣΥΣ. Η αναθεώρηση έγινε πέρσι, την εγκρίναμε, πέρασε δηλαδή από μας. Είπατε ότι ως το τέλος του 20 θα πρέπει τα τεχνικά εργαλεία να διατηθούν στα κράτη-μέλη. Είναι όμως σχεδόν έτοιμα, είναι η ερώτησή μου. Έχει γίνει απαραίτητη δουλειά και από τα κατημέλια. Και μια ακόμη ερώτηση, να με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Πήγα στην έδρα σας στο Στρασβούργο πριν από κάμποσο καιρό για όλα τα νέα συστήματα που αναπτύσσετε. Έχω να πω ότι δεν είναι και πολύ σύγχρονο το μέρο, ούτε πολύ ε, εντυπωσιακό. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για την Ιουλίσσα, μιλάμε για πολλές προκλήσεις, πολλά καθήκοντα, προστασία δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων. Πρέπει να οργανώσουμε ε, όλες τις διάφορες βάσεις δεδομένων, μιλάμε για διαλειτουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τα διάφορα συστήματα των κρατών μελών. Ε, πρέπει να εντοπίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα η Ιουλίσα δεν είναι από τις μεγαλύτερες υπηρεσίε που έχουμε. Οπότε το ερώτημά μου είναι μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις παλές και τις νέες προκλήσεις ε, με τις δυνατότητες, ε, τα μέσα που έχετε ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα ε, και χρηματικό και οικονομικό και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα προστασίας δεδομένων δυσκολεύεστε να βρείτε το κατάλληλο προσωπικό για όλα αυτά τα καθήκοντα ή τα καταφέρνετε. Ευχαριστώ κυρία Κελέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Κάρκοφ ε, και σας και, το, και την ομάδα σας για το έργο σας στα πλαίσια της EU Lisa. Το, το ερώτημά μου συμπίπτει με αυτό της κυρία Σίπερ. Σίπελ, μπορείτε να μας πείτε για τον προπολογισμό, αρκεί ο προπολογισμό ε, μετά τις νέες εξελίξεις και τις νέες πληροφορίες στις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσετε, πρέπει να εξεργαστείτε, εν Επίσης η κυρία Χέντριξον, υπουργό δικαιοσύνη Δικαιοσύνης ε, της Φιλανδικής Προεδρίας, μας είπε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ασχοληθείτε και με πληροφορίες που έχουν να κάνουν ε, στις, ε, με τις μεταφορές, τις μετακινήσεις ε, με πλοίο και με τρένο. Είχε ξεκινήσει όλο κάτι τέτοιο. Η κυρία Ντάλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε φαντάζομαι ότι το βασικό μου ερώτημα έχει να κάνει με ε, τα ζητήματα που, κρύβονται πίσω από τα, τις προσπάθειες αυτές. Η διαλειτουργικότητα, ε, η απειλή για την, εστερική, ασφάλεια, νέες προκλήσεις, η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων αναφέρει ότι όλο και πιο συχνά συνδέουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης με την ε, ασφάλεια ε, και το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο διότι τι λέμε τελικά η μετανάστευση είναι μια απειλή για την ασφάλεια οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα, αυτά τα μονολυθικά συστήματα ε, πληροφοριών που είναι μια απειλή στην ιδιωτική ζωή και στη θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί γιατί συμβαίνει αυτό, ποιο στοιχείο αποδεικνύει αυτή τη στιγμή ότι η μετανάστευση αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και ότι αυτοί οι μηχανισμοί καθιστούν την Ευρώπη πιο ασφαλή. Τι ε, αιτιολογεί αυτό το επιχείρημα, αυτό το συμπέρασμα, διότι για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να το αιτιολογεί. Δεν είναι βέβαια προσωπική επίθεση προς εσά, αλλά για μένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ε, ότι αυτή είναι η βάση αιτιολόγησης ε, των ε, ε, εργασιών σας, μια βάση που είναι λανθασμένη. Αντί να σταματήσουμε να παραμβαίνουμε στη Μέση Ανατολή και να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για να ασφαλίσει οι άνθρωποι αυτές τις χώρες τους, χωρίς να χρειάζεται να κλείνουμε τα σύνορά μας. Λοιπόν, ωραία, σε λίγο θα περάσουμε το χρόνο, οπότε προσπαθήστε να είστε σύντομος, όσο γίνεται πιο σύντομος. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι, συγγνώμη, ξέχασα κάποιον. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να θέσω για την πρόσβαση σε βάση δεδομένων. Ε, αναφερθήκατε στην περίπτωση hackers που έχουν πρόσβαση σε βάση δεδομένων. Τι γίνεται όμως με την επίσημη πρόσβαση. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, έχει ένα αντίγραφο του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν και το χρησιμοποίησε καταχρηστικά από ό,τι μάθαμε. Υπάρχει σε τεχνικό επίπεδο κάποιο μέτρο για να προλάβουμε τα αντίγραφα, την αντιγραφή της βάσης δεδομένων και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση από επισήμους από στη στην Γερμανία, είχαν πολλές περιπτώσεις όπου αστυνομικοί είχαν πρόσβαση σε βάση δεδομένων για ιδιωτικού λόγους, από περιέργεια, για να δουν Παραδείγματο χάρη, ε, τι κάνει κάποια προσωπικότητα ή κάποια διασημότητα. Έχετε κάνει κάτι για να προλάβετε την καταχρηστική πρόσβαση εξωματούχων, να του ζητείτε, παραδείγματο χάρη, ε, να αιτιολογήσουν την πρόσβασή του. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Θα τα απαντήσω με τη σειρά. Για τις εκκρεμείς προτάσεις της ΛΥΜΠ, για τις τροπολογίες της, του αίτιας Eurodac και το καθεξής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιες τοπολογίες ζητούν αλλαγές και στο ΕΤΙΑΣ και στο ΙΕΣ τους σχετικούς κανονισμούς για την ε, αναδρομική διαλειτουργικότητα. Χρειάζονται οι τροπολογίες αυτές για να εφαρμοστεί σωστά το ΕΤΙΑΣ, η διαλειτουργικότητα και το ΙΕΣ, όπως είχαν σχεδιαστεί. Οπότε, εάν δεν ολοκληρωθεί η συζήτηση για τι τροπολογίε αυτές, ε, υπάρχει κίνδυνο. να καθυστερήσουμε το ΙΕΣ e να διατεθεί πρώτη φορά στα τέλη του 20 και μετά από ένα χρόνο τα επόμενα δύο. Το ΙΤΕΑΣ e και το διαλειτουργικότητα. Πρέπει να ολοκληρωθούν λοιπόν οι προτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Έχει να κάνει και με την ικανότητα του οργανισμού. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και τα έχουμε πει. Το ίδιο και για το, την ε, αναθεώρηση, την αναδιατύπωση Eurodac. Το Eurodac και το VAS είναι καθοριστική σημασία ε, τμήματα του αρχιτεκτονήματος για τη διαλειτουργικότητα. Όσο πιο πολύ καθυστερούμε, τόσο πιο πολύ θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Τα κάτι μέλη είναι έτοιμα για την υλοποίηση. Ε, ο οργανισμός συνεργάζεται πολύ στενά και παρακολουθεί την υλοποίηση στα περισσότερα κάτι μέλη είναι στο σωστό σημείο για τη διαλειτουργικότητα και τα σημεία εξόδου και εισόδου. Κάποια κάτι μέλη αντιμετωπίζουν όντω δυσχέρειε, αλλά μαζί με την Επιτροπή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να τα υποστηρίξουμε. Για να ξαναμπούν στο σωστό ρυθμό. έδρα του οργανισμού στο Στρασβούργο. Μόλις ε, ολοκληρώσαμε το πρώτο παράρτημα εκεί. Δεν έχουμε όμως αρκετούς πόρους. Γι' αυτό το είπα και ξεκάθαρα. Μια από τις δυσκολίες του οργανισμού στο εγγύς μέλλον είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο